Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε. Το επόμενο θέμα είναι η αναθεώρηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών ενεργείων μεταφορών. Συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ειδήσει ο κύριος Μπαχ. Πρώτα θα πάρει το λόγο ο κύριος Μπαχ μετά ο εισηγητής ΙΜΚΟ, ο κύριος Μάια, νομίζω, μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά η προσκεκλημένοι μας. Θα αρχίσει λοιπόν ο George. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα δικαιώματα των επιβατών ε, εναερίων μεταφορών είναι πολύ σημαντικό τα δικαιώματα των επιβατών γενικά είναι για όλες ε, τις ε, μορφές μεταφορών και συγκοινωνιών πολύ σημαντικό θέμα. Δεν αφορά μόνο τους επιβάτες, αλλά συνολικά τον πληθυσμό, αλλά και τον κλάδο. Και όπως βλέπετε, βλέπετε λοιπόν ότι αφορά τους διάφορους φορείς του κλάδου, τις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια Όλοι πρέπει να τηρήσουν και στο μέλλον, να τηρούν τους κανόνες για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Τι περιμένουν από εμά με βάση και την ομοθεσία αλλά και την ομολογία. Στην ομοθεσία λοιπόν του 2004 υπήρχαν ασάφειες, υπήρχαν κενά. Το νέο νομοθέτημα δεν πρέπει να ξανακάνει τα ίδια σφάλματα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να χρειαστεί να ασχοληθούν τα δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συγκεκριμένα για να διευκρινίσουν ασάφειες. Η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται και στην ομολογία σε μεγάλο βαθμό συμμορφούνται αλλά το να έχει κανείς δικαιώματα είναι ένα πράγμα το να απολαμβάνει των δικαιωμάτων αυτών είναι κάτι διαφορετικό η Κομισιόν λοιπόν προσπαθεί να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή και μεταγραφή της νομοθεσίας. Πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικές εποπτικές αρχές και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Πάει προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρόταση. Όταν είναι ενημερωμένοι οι επιβάτες, όταν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές, όταν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους πριν, κατά και μετά την πτήση και όταν γνωρίζουν συγκεκριμένα πού πρέπει να απευθυνθούν για να απαιτήσουν την ε, τήρηση των δικαιωμάτων τους, θα έχουμε επιτύχει ουσιώδη πρόοδο. Κάποια σημεία που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και εμένα βεβαίως αλλά και το ΕΛΚ συνολικά είναι να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις, ιδιαίτερα οι περιπτώσεις Sturgeon Νέλσον αυτός ο κανόνας των τριών ωρών. Πρέπει να το συζητήσουμε Αυτό τον κανόνα. Πολύ σημαντικό είναι οι έκτακτες περιπτώσεις, οι έκτακτες περιστάσεις. Η Κομισιόν ε, ε, προτείνει ένα κατάλογο. Καλός είναι αυτός ο κατάλογος των έκτακτων περιστάσεων, αλλά χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες ε, τροποποιήσεις και να γίνουν πιο δεσμευτικές ρυθμίσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της πολιτικής ε, όταν δεν εμφανίζεται ο επιβάτης, το no-show. Νομίζω ότι οι προτάσεις της Κομισιόν ε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ε, υπέρ των συμφερόντων των πελατών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, αναφέρεται αλλά και εδώ θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και επίσης η καθυστέρηση κατά την άφηση. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα με τις ανταποκρίσεις. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε γιατί σχεδίζεται και με τις ε, συνεργασίες αεροπορικών εταιριών. Κάτι άλλο σημαντικό για τους επιβάτες. Οι χειραποσκευές. Δεν συμφωνώ στο σημείο αυτό με την πρόταση της Κομισιόν. Αυτή η δυνατότητα να αποφασίζουν οι εταιρείε μόνες τους για το πόσες ε, χειραποσκευές θα επιτρέπουν. Πρέπει να υπάρχει ε, ισχυρότερη ρύθμιση. Ε, να λάβουμε υπόψη και την έκθεση Taylor και τη δική μου, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας που περιέχουν την επιχειρηματολογία μας. Ένα άλλο θέμα σε θέματα ε, πτωχεύσεως ε, αερομεταφορέων. Κατά τη γνώμη μου, η ανακοίνωση της Κομισιόν είναι υπερβολικά ήπια, δεν είναι αρκετά σαφής. Ήδη το 2009 η Κομισιόν είχε, εκφρα... ή, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει περισσότερη ευκρίνεια, σα, σαφήνεια δηλαδή, για το τι θα γίνεται σε περιπτώσεις ε, πτωχεύσεων. Χθες ε, κάναμε μια συζήτηση με τους Κιώδης, ε, συζητήσαμε, να, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα του κλάδου. Οπωσδήποτε ένα θέμα που δεν πρέπει να το υποτιμούμε λόγω και της κρίσης. Σήμερα, σε αυτή την ακρόαση, για την οποία ευχαριστώ και τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για αυτά που θα μας πούν. Προσβλέπω σε αυτά που θα μας πούν για να λάβουμε επιπλέον ε, πληροφόρηση και προσβλέπω και στην περαιτέρω συζήτηση και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιερ, Ίμκο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό στην ΙΜΚΟ. Εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών δηλαδή. Ο κανονισμός αυτός λέγεται μέτρα αποζημίωσης και στήριξης των επιβατών. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Η Επιτροπή μας έχει προτείνει λοιπόν με βάση το άρθρο 50 να υπάρξει κοινή συζήτηση αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία του άρθρου 49 συν. Θέλω να υπάρξει συμφωνία, όπως προτείνω, μεταξύ των δύο επιτροπών, ούτω ώστε να συνεργαστούμε πολύ μαζί τους, να συμμετάσχουμε προσκεκλημένοι και στον τριμερή διάλογο. Διότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, το αποδίδουμε μεγάλη σημασία, έχουμε πολλή πείρα, για παράδειγμα, πληροφόρηση των καταναλωτών και θέλουμε και εδώ να συμπεριληφθεί με πολύ βάρος. Για παράδειγμα, το θέμα η καθυστέρηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για τον καταναλωτή αν είναι τρεις ή πέντε ώρες το κατόφλι αποζημίωσης. 100 ευρώ ανανύχτα ναι, αλλά ε, αυτό έχει να κάνει με το πού θα πρέπει να διανυκτερεύσει ο καταναλωτής. Γιατί υπάρχουν μέρη όπου χρειάζονται πάνω από 100 ευρώ για να μπορέσει να διανυκτερεύσει κανείς. Πρέπει να δούμε αυτές τις λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, προσβλέπω και εγώ στην ακρόαση και φυσικά θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, δεν είναι ακριβώς ακρόαση, είναι ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Να το διευκρινίσω. Από την Επιτροπή. Ο Jean-Luc Coulson, τμήματάρχης για δικαιώματα των επιβατών. Δέκα λεπτά αυστηρά. Θα ακούσετε το σφυρί μου αν τα υπερβείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε ότι είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο κανονισμός 261. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Και γιατί. Επειδή λόγω τεσσάρων θεμάτων. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν γκρίζες ζώνες ε, ρυθμιστικές ε, που έχουν οδηγήσει σε πολλές προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεύτερον διότι τα άτομα επιβάτες προσκρούν σε δυσκολίες όταν προσπαθούν να αξιώσουν τα δικαιώματά τους και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Και επειδή η εποπτεία και η επιβολή έχει αποδυναμωθεί από τα όργανα επιβολής του νόμου και τέταρτον διότι υπάρχει κόστος δυσανάλογο για τους αερομεταφορείς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων. Αυτοί είναι οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους η Κομισιό ε, θέλει θέλησε να κάνει μια πρόταση να διευκρινίσουμε τις γκρίζες ζώνες, οι κυρώσεις και η υποπτία να έχουν οι επιβάτες στα εργαλεία τα μέσα να αξιώσουν τα δικαιώματά τους και επίσης λαμβάνουμε υπόψη τις πρακτικές και οικονομικές συνέπειες για τον κλάδο των αερομεταφορέων. Θα ήθελα να επανέλθω σε καθένα από αυτά τα σημεία. Διευκρίνηση των κρίζων ζωνών κάνουμε πολλά σχετικά με τις έκτακτες περιπτώσεις. Έχουμε έναν ορισμό σαφή στον κανονισμό, περιλαμβάνουμε την ομολογία και καμιά φορά είμαστε ακόμα πιο αυστηροί από την ομολογία. Έχουμε επίσης το θέμα του αναπρογραμματισμού. Ο αναπρογραμματισμός, η αλλαγή στον προγραμματισμό των δρομολογίων δεν έχει διευκρινιστεί ούτω ώστε να αποφευθούν οι αποζημιώσεις και να μην θεωρούνται οι ακυρώσεις ακυρώσεις. Πρέπει επίσης ε, να δούμε ε, σε περιπτώσεις ε, διεκπαιρέωσης τι γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχουν προθεσμίες. Ξεχωρίζουμε την λειτουργία της παρακολούθησης και των κυρώσεων και το θέμα της διεκπαιρέωσης των καταγγελιών από την άλλη πλευρά. Όσον αφορά τις, ε, τα εθνικά όργανα επιβολής, θέλουμε ένα δίκτυο άτυπο των εθνικών οργάνων. Θα ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και τις αναφορές από τα όργανα αυτά. Το πεδίο της επιβολής θα περιλαμβάνει επίσης και τα θέματα αποσκευών. Και τελευταίο θέμα, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό όσον αφορά το κόστος, θα πρέπει το κόστος για τις αερομεταφορές να είναι ελεγχόμενο και για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το στόχο της, του κανονισμού αλλάξαμε μερικές, μερικά τμήματα της πρότασης, δηλαδή δεν θα έχουμε το θέμα των τριών ωρών για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων, οι τρεις ώρες θα γίνουν πέντε ώρες. Υπάρχουν μερικές κριτικές σχετικά με την πρόταση αυτή. Μερικοί θέλουν ο κανονισμός να είναι πάρα πολύ σαφής, αλλά τώρα λένε ότι είναι ιδιαίτερα λεπτομερής και περιλαμβάνει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεύτερον, από τους αερομεταφορείς ακούμε πολλές κριτικές σε σχέση ε, με τις χαμένες ανταποκρίσεις. Υπάρχει μια απειλή, λένε, ότι αυτό ε, θα οδηγήσει σε συμφωνίες. Ε, το κείμενο ήδη καλύπτει τις ανταποκρίσεις όπως έχει επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στην περίπτωση ε, C11 Focus. Και η πρότασή μας απλώς διευκρινίζει πως η φροντίδα ε, και η αποζημίωση θα παρέχονται και από ποιον. Οι αερομεταφορείς είναι ελεύθεροι να διευκρινίσουν πώς η επιβάρυνση θα κατανεμηθεί μεταξύ τους. Δεν εισάγουμε τίποτα που να μην υπάρχει ήδη σήμερα. Απλώς διευκρινίζουμε την κατάσταση. Η αποζημίωση για μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 5 ωρών και όχι άνω των 3 ωρών που προβλέπονται από την ομολογία θεωρείται ως μείωση των δικαιωμάτων των επιβατών. Ας είμαστε σαφείς ως προς το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστηριό δεν είχε άλλη επιλογή από το να θεωρήσει τρεις ώρες με βάση τον ορισμό της καθαρά νομικίστικης ανάγνωσης της ισχύουσας ε, ε, νομοθεσίας. Δεν χρειάζεται οικονομική αξιολόγηση συνδυασμένη με αυστηρό ορισμό των εκτάκτων περιστάσεων που προτείνουμε. Ένα κατώτατο όριο ε, των τριών ωρών θα αυξήσει δυσανάλογα το κόστος για τους αερομεταφορείς και θα παρακινήσει τους αερομεταφορείς να ακυρώνουν τις πτήσεις. Τέσσερα, το θέμα της επαναδρομολόγησης η επαναδρομολόγηση με τον ίδιο αερομεταφορέα εντός 12 αερών είναι τώρα κάτι το υποχρεωτικό, αλλά δεχόμαστε κριτικές τόσο από τους αερομεταφορείς που παραπονούνται ότι 12 ώρες είναι πολύ λίγο και οι επιβάτες που παραπονούνται ότι 12 ώρες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήμουν χτες στην Οικονομική και Κοινωνική Επίτροπη και όλοι λέγανε ότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, προτείνουμε 12 ώρες, διότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ε, διότι θα ξέρει έτσι ο επιβάτης από ε, ποια στιγμή μπορεί να απαιτήσει επανοδρομολόγηση, αλλαγή δρομολογίου με όλες, με όλες τα, τις παροχές φοβούνται οι αερομεταφορείς ότι αυτοί οι κανονισμοί θα αποθαρρύνουν τους επιβάτες να κάνουν αγορές στα, στους αερολιμένες. Βεβαίως αυτός ο κανόνας ισχύει από ορισμένους ορμεταφορείς από την άποψη των επιβατών και όχι των επιχειρήσεων. Το βασικό πρόβλημα από την πλευρά των επιβατών είναι ότι υπάρχει σύγχυση το τι επιτρέπεται να πάρουν πάνω στο αεροπλάνο. Και εμείς προτείνουμε περισσότερη διαφάνεια ως προς το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σας πω και πάλι ότι η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση ε, των ε, νομοθετών κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Κόλσον και τώρα ε, θα ασχοληθούμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι αερολιμένες, οι αερομεταφορείς και οι καταναλωτές και πρώτα δέκα λεπτά είναι από το Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων ο κύριος Μόργαν Φούλξα, ε, ε, υποδιευθυντής. Έχετε 10 λεπτά για να μας κάνετε την παρουσίασή σας και μετά θα έχουν οι αερομεταφορείς 5 λεπτά ο καθένας, διότι έχουμε περισσότερες ενώσεις αερομεταφορέων. Έχετε λοιπόν 5 λεπτά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού που μας δίνει εδώ την ευκαιρία να λάβουμε τον λόγο και ελπίζω να συμβάλλω θετικά στην εργασία αυτής της Επιτροπής. Εκπροσωπούμε 178 178 σε 46 χώρες και μαζί αντιπροσωπεύουν 90% της κυκλοφορίας ε, στα ε, και αντιπροσωπεύουμε 8 επίσης ε, ενώσεις εθνικών αερολιμένων. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι περισσότερο ένα πρόβλημα έλλειψης επιβολής και τήρησης των κανονισμών και αυτό αναγνωρίζεται στο άρθρο 16.2 ε, της αιτιολογικής, ε, του αιτιολογικού ε, μνημονίου και τα στοιχεία τα νομικά που απαιτούνται στην πρόταση 3.3.1.2. Θα πρέπει τα δικαιώματα να τηρούνται. επίση η έλλειψη εφαρμογής αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες ερμηνεύουν διαφορετικά τον κανονισμό 261 και το τι είναι μέσα στο πεδίο εφαρμογής ή εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 261. Η ερμηνεία λοιπόν είναι διαφορετική ανάλογα αν πρόκειται για αερομεταφορείς ή για άλλους. Έχουμε λοιπόν υποστήριξη πέραν των νομικών υποχρεώσεων σε καθυλωμένους επιβάτες. Έχουμε ε, περίπου ε, πάρα πολλούς επιβάτες που ε, ταξιδεύουν χωρίς βίζα, που έχουν χωριστά εισιτήρια και χάνουν ένα τμήμα, ένα μέρος της πτήσης τους. Όταν είχαμε την κρίση του νέφους από το ηφαίστειο, είχαμε διακοπές, διαταραχές και στο Σκύπολ και επίσης και χρειάστηκε να παρασχεθεί γιατρική φροντίδα, ειδική φροντίδα στα παιδιά και ε, το κόστος ε, για τους αερομεταφορείς ήταν της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό ε, είναι 50 ευρώ ανά ημέρα ανά επιβάτη. Λοιπόν, στην πρόταση θέλουμε να διευκρινίσουμε καλύτερα την εφαρμογή των δικαιωμάτων. Βεβαίως, οι αερομεταφορές έχουν την πρωταρχική ευθύνη απέναντι στους επιβάτες. Πρέπει να διευκρινίζουν τις έκτακτες περιστάσεις. Υπήρξε βελτίωση της νομοθεσίας, παραμπτός χάρη, το δικαίωμα να διορθώνονται τα ονόματα που δεν έχουν γραφεί καλά ορθογραφικά, να απλουστευτεί η διεκπαιρέωση των καταγγελιών και να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών ε, οργάνων. Επίσης ε, δεν αναφέρει τίποτα ο κανονισμός για την ανάγκη των αερομεταφορέων να έχουν ένα αντιπρόσωπο τοπικό για χαμένες αποσκευές θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή στο άρθρο 14, ούτω ώστε οι αερομεταφορεί να έχουν μια επαφή, ένα άτομο επαφή στα αεροδρόμια, ίσως όχι δικό του υπάλληλο, αλλά κάποιον όταν το χάρη αρνείται σε κάποιον η επιβίβαση, όταν υπάρχουν αιματεώσει πτήσεων, οι μεγάλε καθυστερήσει σε σχέση με την φροντίδα, την επιστροφή χρημάτων, την αναδρομολόγηση, τον ανασχεδιασμό, ε, κράτηση νέων εισιτηρίων. Όλα αυτά έχουν αναφερθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο Υπάρχουν επίσης νέες υποχρεώσεις για τους αερολιμένες. Δεν υπάρχει τυπική ε, υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Η αρρωγή παρέχεται σε θελοντική βάση. Υπάρχουν δύο μεγάλες υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης ε, στα αεροδρόμια άνω των 3 εκατομμυρίων ατόμων και επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 υπάρχουν υποχρεώσεις ενημέρωσης. Πολλές αεροπορικές εταιρείε έχουν ίδια σχέδια εκτάκτου ανάγκης, δεν είναι αυτό πρόβλημα. Χρειάζονται απλώς μερικές διευκρινήσεις στο άρθρο 5.5. Τι ποιο γεγονός πυροδοτεί την ανάγκη να εφαρμοστούν σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Ως προς την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 14, πολύ αερολιμένες στην περιοχή όπου γίνεται το check-in και η επιβίβαση παρέχουν πληροφορίες, αλλά το άρθρο 14 προχωράει ακόμα περισσότερο και λέει ότι οι, τα, αερολιμένες θα πρέπει να ενημερώνονται για την ακύρωση της πτήσεως ε, βεβαίως τα αεροδρόμια εξαρτώνται από τους αερομεταφορείς για να μπορούν να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε επίσης το δικαίωμα επανόρθωσης, ε, άρθρο 13, το θέμα το τι επιτρέπεται ως προς τις αποσκευές, τις καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο, προς τον ρόλο και την ευθύνη των διαφόρων ε, συμμετεχόντων. Έχουμε επίσης τον ορισμό και τον ρόλο του, της διεύθυνσης του και παρόλο που δεν υπάρχει στον κανονισμό τίθενται ορισμένα ερωτήματα και θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε τα πράγματα διότι οι αερολιμένες δεν μπορούν να ελέγξουν τους διάφορους πρωταγωνιστές, μπορούν να τους συντονίζουν, να τους ελέγχουν. Επίσης πρόκειται για μια συνεργατική προσπάθεια σε έκτακτη ανάγκη. Επίσης ε, τα αεροδρόμια ε, κάτω των τριών εκατομμυρίων. Επίσης πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την ευθύνη τους. Υπάρχει επίσης μια εναλλακτική γλώσσα ε, όχι στον κανονισμό αλλά στον τον τωρινό κανονισμό, αλλά στον κανονισμό 1108 του 2009 σχετικά με την αεροπορική κυκλοφορία, σχετικά με τους οργανισμούς, έχουμε τον ορισμός που έχουμε στο άρθρο 5.5 μας λέει για τα δικαιώματα επιβολής, τα αερολιμένες δεν μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις. Η ικανότητα ε, τήρησης ε, ε, και επιβολής κυρώσεων είναι ευθύνη και υποχρέωση των εθνικών οργάνων επιβολής του κανονισμού. Θα ήθελα να μιλήσω για το άρθρο 6 σχετικά ε, με, την, ε, με τις συνδέσεις τις περιφερειακές. Ήρθαμε σε επαφή με περιφερειακούς αερομεταφορείς. Υπάρχει μια δυσαναλογία στο άρθρο αυτό ε, σχετικά με τις, με, τους με τις περιφερειακές πτήσεις. Υπάρχουν, μερικοί, υπάρχουν μερικές συμφωνίες μεταξύ ορισμένων γραμμών και αερομεταφορέων ότι να αναγκάζονται οι επιβάτες να αγοράζουν ξεχωριστά χωριστά εισιτήρια, ε, να, να παίρνουν τις αποσκευές τους, να χρειάζεται και πάλι να ελεγχθούν και να παραδοθούν. Όλα αυτά, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, ε, θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα, διότι αυτό έχει ε, συνέπειες πάνω στις περιφερειακούς αερολιμένες και επίσης ε, ε, δημιουργείται συμφόρηση, ε, ανώφελη άχρηστη συμφόρηση σε ορισμένους κόμβους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει καλή προστασία των επιβατών. Έχουμε το θέμα του κανόνα της μιας αποσκευής που αναφέρεται στον κανονισμό 2027 ε, και έχουμε περιοριστικές πολιτικές ε, τα πρόσφατα χρόνια σχετικά ε, με τα, τις αποσκευές που μπορεί κανείς να έχει στο θάλαμο των επιβατών, να παίρνει μαζί του. Θα υπάρχει ελευθερία για τους αερομεταφορείς, για τις αποσκευές που μπορεί ο επιβάτης να πάρει μαζί τους, ενώ υπάρχει καλή ενημέρωση. Νομίζω ότι αυτός ο κανόνας έχει μεγάλες συνέπειες πάνω στους επιβάτες ε, και βεβαίως ε, αμφισβητεί μια πρακτική 60 ετών, οδηγεί σε σύγχυση διότι μπορεί να ποικίλουν οι κανόνες ακόμα και ε, στα πλαίσια ενός ιδίου αερομεταφορέα. Επίσης μειώνει την ελευθερία επιλογής ε, για τους επιβάτες όταν κάνουν αγορές στο αεροδρόμιο. Επίσης έχει επιπτώσεις πάνω στους αερολιμένες, απειλεί το οικονομικό μοντέλο και την βιωσιμότητα των αερολιμένων αερολιμένων. Επίσης ε, έχουμε τα αεροδρόμια που είχαν μεγάλες ζημίες και επίσης 65% ε, στα αεροδρόμια κάτω του ενός εκατομμυρίου επιβατών έχουμε μη αεροναυτικά έσοδα τα οποία είναι 41% των εσόδων των αερολιμένων και καμιά φορά μέχρι 70%. Επίσης μειώνεται το εισόδημα το εμπορικό και οδηγεί σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους αερολιμένες. Έχει κάνει έκκληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και εμείς υποστηρίζουμε την αλλαγή στην πρόταση για την προστασία των επιβατών εναντίον των υπερβολικά περιοριστικών μέτρων και να μπορούν να έχουν μαζί τους αποσκευές για να μπορούν να κάνουν και αγορές στα καταστήματα των αερολιμένων. Uh, Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Έχουμε τέσσερις ενώσεις αερομεταφορέων θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Μονίκ Ντεσμέτ, Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ευρώπη της ΙΑΤΑ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών διότι προσκάλεσε την ΙΑΤΑ σε αυτήν την ε, ανταλλαγή απόψεων. Εκπροσωπούμε 240 αερομεταφορείς, 60 εκ των οποίων εδράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων των 32 εταιριών της AEA. Οι υπόλοιπε πετάνε από και προς την Ευρώπη, επομένως επηρεάζονται από τον σχετικό κανονισμό και την αναθεώρησή του. Μπορέσαμε, πέρα από το ότι έχουμε μέλη από όλες τις αεροπορικές εταιρείες που ακολουθούν όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, είμαστε περήφανοι λοιπόν που μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις όχι μόνο της ΙΑΤΑ και της ΑΕΑ, αλλά και της ΕΛΦΑΑ, της ΕΡΑ και της ΙΑΚΑ, ε, εκπρόσωποι των οποίων θα πάρουν το λόγο αργότερα και θα σχολιάσουν και αυτοί τις ανησυχίες που έχουμε όλοι για την αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι είναι καλό πράγμα η αναθεώρηση. Ο κανονισμός 261 περιλαμβάνει γκριζε ζώνες, κάτι το οποίο έχουν επισημάνει πολλές δικαστικές αποφάσεις. Από την αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν γνωρίζουμε ότι έτσι όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή το κόστος είναι μεγάλο και αποθαρρύνεται η βούληση για συμμόρφωση με το κανονισμό. Θέλουμε λοιπόν την αναθεώρηση του κανονισμού, εάν διευκρινίσει τις διατάξεις, εάν βελτιώσει την αρμονισμένη εφαρμογή και αν ε, προσδώσει πραγματικά πραγματικά επιπρόσθετα δικαιώματα στους επιβάτες. Πραγματικά επιπρόσθετα ε, δικαιώματα. Φροντίδα για όλους τους ε, επιβάτες, ε, δύο ώρες μετά το πρόβλημα, σε αρχικό στάδιο δηλαδή, καλύτερη πληροφόρηση στους επιβάτες το συντομότερο δυνατόν, στηρίζουμε την αναθεώρηση εκεί όπου βρίσκει ένα νέο σημείο ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων επιβατών και των υποχρεώσεων των αερομεταφορέων. Η αλλαγή του σημείου ισορροπίας είναι ακριβώς και ο πυρήνας του ζητήματος. Η καθυστερημένη αντιστάθμιση ή αποζημίωση ε, το trigger point. Η Κομισιόν το επισημαίνει και λέει ότι αν υπάρχει κάποιο ε, πρόβλημα, σε κάθε περίπτωση κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι καθυστερήσεις ε, σημαίνουν ένα υψηλό λειτουργικό κόστος για τους αερομεταφορείς. Οι εταιρείε κάνουν το παν για να μειώσουν τις καθυστερήσεις για να μην έχουν ε, υψηλό κόστος που θα πρέπει να αναλάβουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν περιλήφθη η υποχρέωση αποζημίωσης για καθυστέρηση στην τωρινή αναθεώρηση, γιατί έχει ήδη περιληφθεί αυτό στο 261 ούτω ή άλλω. Μπορεί οι εταιρείε να επιλέξουν να ακυρώσουν την πτήση παρά να την εκτελέσουν υπερβολικά καθυστερημένη. Η Κομισιόν τελικά κατάλαβε ότι κάλιο αργά παρά ποτέ και με το trigger point στο σημείο πυροδότηση, αν θέλετε, ε, μπορούν οι εταιρείε να λύσουν το πρόβλημα Καλωσορίζουμε επίσης το γεγονός ότι φάνηκε από τον έφος ηφαιστιακή τέφρας ότι δεν φταίνε μόνο οι αεροπορικές εταιρείες για την παροχή βοήθειας και στέγασης σε περίπτωση προβλήματος που είναι μαζικό και που ε, ξεπερνά ε, τις δυνατότητές τους. Ερχόμαστε τώρα σε αυτά που δεν μπορούμε να δεχθούμε γιατί δημιουργούν ψευδή επιβατικά δικαιώματα. Θα θέλαμε οι προτάσεις αυτές αυτές να μην υιοθετηθούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι ποιο. Αναμφίβολα η ασφάλεια και είναι και θα πρέπει να παραμένει υπαριθμόν ένα προτεραιότητα καταστάσεις όμως που δεν μπορεί να ελέγξει η εταιρεία τελικά ε, θέτουν ένα αμφιβόλο την ασφάλεια της πτήσης και θα πρέπει να θεωρούνται ως ε, κατεξαίρεση ε, περιπτώσεις και να μην επιβάλλεται στον αερομεταφορέα να πληρώσει κατά αποκοπήν ποσό αποζημίωσης ο αερομεταφορέας θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση διότι υποχρεώνει έναν επιβάτη να συμμορφούνται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον άβλο που επέλεξε ο επιβάτης να αγοράσει. Ορισμένοι επιβάτες δεν γνωρίζουν κάτι που θα έπρεπε. Και όντως οι συμβατικές υποχρεώσεις θα πρέπει να ε, γίνουν πιο σαφείς. Ότι δηλαδή ε, θα πρέπει τα εισιτήρια να χρησιμοποιούνται όλα τους τα κομμάτια. Δεν μπορώ να επεκταθώ τώρα στις πολιτικές τιμολόγησης των εταιριών. Ωστόσο το σημείο κίνησης ενός ταξιδιού είναι πολύ σημαντικό για τον καθορισμό της τιμής αυτού του εισιτηρίου όλες αυτές τις διαδρομές. Σχετίζονται όλα αυτά με την ελεύθερη αγορά. Το να απαγορεύσουμε στις εταιρείε να προβλέπουν κάτι τέτοιο είναι κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά τους ναύλους και μάλιστα πολύ. Οι συνθήκες ε, υπό τις οποίες θα παγορευτεί ε, η πολιτική του no-show όταν δεν εμφανίζεται ο επιβάτης ε, θα δώσουν το δικαίωμα στους επιβάτες να κοροϊδεύουν το εισαγωγικών της επιχειρήσεις και να μην συμμορφούνται με το δικό τους κομμάτι. Ε, δίδεται έτσι το κίνητρο για τις εταιρείες να κάνουν overbooking, να έχουν υπεράριθμες κρατήσεις, κάτι το οποίο θα είναι επί παραβάση του κανονισμού 261. Εναλλακτική των υπεράριθμων πτήσεων είναι να πετάμε με κενά καθίσματα, το οποίο δεν είναι καλό για το περιβάλλον, εάν απαγορευτεί η πολιτική που έχουμε για το no-show. Ε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, και τώρα με τις καταλεκτικές μου παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή σε αυτά που θα πει ο επόμενος ομιλητής. Το τρίτο σημαντικό σημείο δηλαδή. Κάτι το οποίο θα ε, οδηγήσει σε ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Το θέμα του τελικού προορισμού είναι σημαντικό για όλους, αλλά θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κατατόπους περιφέρειες. Και θα δώσω το λόγο στον Σάιμον Μακναμάρα, ε, συνάδελφό μου από την ΕΡΑ την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακών Αερομεταφορέων. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάιμον Μακταμάρα από την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αερομεταφορέων. Δική μου είναι η συνεδρίαση, εγώ προεδρεύω. Είναι Γενικός Διευθυντής, έχετε πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Καλησπέρα σε όλους. Και εμεί εκτιμούμε ιδιαίτερο το γεγονό ότι μα δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα δημόσια. 51 εταιρείε εκπροσωπούμε, ε, κυρίω αερομεταφορεί ε, με μικρά αεροσκάφη που διανύουν μικρέ αποστάσει και ε, τροφοδοτούμε και τους αεροπορικούς κόμβους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα επανέλθω αργότερα. Βλέπετε κάποια από τα μέλη μας στην οθόνη, κάποια θα τα γνωρίζετε, κάποια θα τα βλέπετε για πρώτη φορά. Όμως πετούν με μικρότερα αεροσκάφη, παρέχουν υπηρεσία από ένα σημείο στο άλλο και έχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε hub fit operation, δηλαδή μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας βασίζεται στο ότι προσφέρουν την ανταπόκριση στις πτήσεις των μεγάλων εταιριών. Γνωρίζετε τη θέση που έχει ο κλάδος ως προς τον κανονισμό 261, προκαλεί σύγχυση και στους, στις εταιρείες και στους καταναλωτές. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η ευκαιρία βελτίωσης του κανονισμού. Ε, καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν γιατί μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε αυτό τον κανονισμό και να το βελτιώσουμε. Και συμφωνώ και με πολλά από αυτά που είπε η Μονίκ. Θέλουμε να προβάλλουμε μια ενωμένη εικόνα εδώ εμείς όλες οι ενώσεις. Ωστόσο θέλω να μιλήσω κυρίως για το θέμα των πτήσεων ανταπόκρισης και έτσι όπως διαπτυπώνεται στο 6α και στο τέλος θα αναφέρω και δύο άλλα ζητήματα. Το σύστημα Hub and Spoke είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας δίνει ανταποκρίσεις από τις κατατόπους περιφερειές στον υπόλοιπο κόσμο. 19.000 πτήσεις εβδομαδιαίως εμφανίζονται σε όλους αυτούς τους ναύλους ε, που εκδίδονται και πολλούνται και ε, διασφαλίζουν τη μεταφορά από τις περιφέρειες στον υπόλοιπο κόσμο. Η ε, αλλαγή για τις πτήσεις ανταπόκρισης έτσι όπως παρουσιάζεται στο 6α είναι πρόβλημα. Ένα παράδειγμα, πτήση από τις νήσους Φαρόε στην μέσω Κοπεχάγης για το Τόκιο. Είναι σημαντική η σχέση μεταξύ των δύο. Σε αυτό το παράδειγμα το πρώτο σκέλος το, του ταξιδιού το προσφέρει ένας περιφερειακός αερομεταφορέας και το δεύτερο σκέλος το προσφέρει ένας αερομεταφορέος δικτύου. Ε, η πρώτη πτήση μπορεί να φτάσει με περίπου 45 λεπτά καθυστέρηση και δυστυχώς ο επιβάτης χάνει την ανταπόκριση για την επόμενη πτήση ε, στο, ε, από Κοπεχάγη για Τόκιο. μία πτήση είναι τη μέρα. Εάν δεν του προσφερθεί ένα διαφορετικό μέσο μεταφοράς, ένα διαφορετικό δρομολόγιο θα πρέπει να, να περιμένει 24 ώρες λόγω μιας καθυστέρησης 45 μόνο λεπτών. Αυτή τη στιγμή ο επιβάτης προστατεύεται ήδη από τη σύμβαση του 99 του Μοντρεάλ. Και έχουμε και πολυμερείς συμφωνίες για ε, ε, διετερικές για την ε, εναέρια κυκλοφορία. Και θα έχουμε λοιπόν ένα δυσαρεστημένο επιβάτη γιατί θα υπάρχει καθυστέρηση, αναμφίβολο αυτό, σίγουρο αυτό, αλλά δεν θα έχουμε έναν απροστάτευτο επιβάτη γιατί ήδη προστατεύεται βάσει των εφιστάμενων κειμένων συμφωνιών και κειμένων. 600 ευρώ είναι η αποζημίωση που καταβάλλεται στον επιβάτη. Είναι δυσανάλογο το κόστος για μια καθυστέρηση 45 λεπτών και τελικά ε, λειτουργεί ως αποθάρρυνση για να εφαρμοστεί η αρχή του hub and spoke. Θα σταματήσει η διεταιρική ε, συμφωνία και συνεργασία τελικά και θα προκληθούν περαιτέρω εμπόδια και ταλαιπωρίες ε, για τον παϊβάτη, ο οποίος θα πρέπει να ξανακάνει check-in τις βαλίτσες από τη στιγμή που θα έχει να συναλλαχθεί με κάθε εταιρεία διαφορετικά και ξεχωριστά. δεν θα θέλουν οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να προσφέρουν ένα ενιαίο εισιτήριο για τη διαδρομή αυτή στην οποία, ε, ε, η οποία εξυπηρετείται από διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικά αεροσκάφη. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Λονδίνο, Ντουμπάι, Μπανκόγκ. Λονδίνο, Μπανκόγκ μέσω Ντουμπάι. Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού διενεργείται ε, χωρίς καθυστέρηση. Το δεύτερο όμως φτάνει αργά η πτήση αυτή, η οποία είναι μη ευρωπαϊκής εταιρείας. Ποιος ο, ευθύνεται. Είναι εκτός πεδίου εφαρμογή της αποζημίωσης ε, το θέμα του δεύτερου σκέλους του ταξιδιού γιατί το εκτελεί ένας αερομεταφορέας που δεν είναι ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και το θέμα του άρθρου 2, το Ι, το κεφαλαίο. Προτείνει η Κομισιόν εκεί όπου μια πτήση αλλάζει διαδρομή, δρομολόγιο, να θεωρείται ακύρωση για οποιοδήποτε λόγο, άρα να ε, ε, συνεπάγεται αυτό αποζημίωση, υποχρέωση ε, καταβολής υποζημίωση. Συγγνώμη, δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη επειδή διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πτήσεων και προτείνουμε μια, ένα διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης, επειδή κάνουμε αυτή την εκτροπή για λόγους ασφάλειας των πτήσεων. Εάν έχετε απορίες ή αν το αφισβητείτε, αναζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εμπειρογνωμόνων και ειδικών περί της ε, ασφάλειας των πτήσεων. Μην πείθετε σε κάτι το οποίο λέει οποιοδήποτε. Ευχαριστώ. Ο Τζον Χάλλον, Γενικός Γραμματέας ε, της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Αερομεταφορέων Χαμηλού Κόστους, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω κάποια θέματα από τον κλάδο των εταιριών χαμηλού κόστου. Συμμερίζομαι τι απόψει που εκφράστηκαν στι προηγούμενε παρουσιάσει. Ακούσαμε το έτοιμά σα, προσπαθήσαμε να συντονίσουμε τι παρουσιάσει μα. Καλωσορίζουμε την αναθεώρηση του κανονισμού. Είναι μια ευκαιρία για να ξανατονίσουμε ότι οι επιβάτες χρειάζονται επαρκή δικαιώματα και να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εμπειρία, ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο λελογισμένη απόδοση του βάρους της αποζημίωσης. Τα τέσσερα σημεία που θέλω να ασχοληθώ είναι το ένα καινούργιο. Τα τρία είναι περαιτέρω επεξήγηση θεμάτων που ήδη αναφέρθηκαν. Πιστεύουμε ότι η χρηματική αποζημίωση για ορισμένες πρακτικές των εταιριών προς το συμφέρον τους ε, αρμόζει να υφίσταται, το αποδεχόμαστε. Τις καθόρισε ο αρχικός κανονισμός πρώτον, ε, επιπλέον επιβεβαιώσεις θέσεων και άρνηση επιβίβασης. Αλλά σε άλλες ε, περιστάσεις που προβλέπεται αποζημίωση, η εταιρεία τιμωρείται όπως και ο επιβάτης και είναι υπερβολική αποζημίωση. Πιστεύουμε ότι πιο δίκαιη, όπως και σε άλλες ε, μορφές μεταφορών, οι οικονομικές κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες ε, του ναύλου. Δείτε περιπτώσεις από το ίντερνετ ε, χθες. 59 ε, ευρώ να πάει κανείς από το Παρίσι στο Μιλάνο με επιστροφή, ενώ σε μια κανονική αεροπορική εταιρεία business θα ήταν 1347 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσουν το ίδιο ποσό και στις δύο περιπτώσεις οι εταιρείες. Άδικο είναι αυτό. Θα προτείναμε αλλιώ για την, ε, το χαμηλότερο ναύλο να είναι ένα ποσοστό ε, του ναύλου με μήνυμου 100 και μάξιμου 250. Έκτακτες περιστάσεις. Η πρόταση της Επιτροπής ε, δεν πηγαίνει αρκετά μακριά για να συνδέσει τις διάφορες πτήσεις που είναι τμήμα του τρόπου λειτουργίας και των δρομολογίων του ίδιου αεροσκάφους θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να επικαλεστούμε έκτακτες περιστάσεις ε, για άλλες πτήσεις που έκανε το ίδιο αεροσκάφος. Αλλιώς στην ουσία ε, μας σωθείτε να ακυρώσουμε πτήσεις. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, γιατί πολλοί θα διαπιστώσουν μετά ότι έχουν πολύ περιορισμένε και καθόλου δυνατότητες αυτά στον προορισμό τους. Αλλαγή δρομολογίου. Βεβαίως, η υποχρέωση να δοθεί άλλο δρομολόγιο θα πρέπει να είναι εντό 24 ώρων, ούτως ώστε να υπάρχουν αλλαγέ λύσει που να εγγυώνται και για την εταιρεία και για τον επιβάτη ότι θα φτάσει στον προορισμό του. Επίσης, κάνουμε έκκληση. Η Επιτροπή έκανε μια προσπάθεια να ε, υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο για τον άβλο που θα πρέπει να πληρωθεί για αυτήν την ε, αλλαγή δρομολογίου θα προτείναμε η μέγιστη, ο μέγιστος ναύλος να μην είναι πάνω από το διπλάσιο του αρχικού ναύλου. Και τέλος, καλύτερη κατανομή του βάρους. Αυτός ήταν ε, ένας από τους στόχους, τους εκπεφρασμένους στόχους όταν ε, ανακοινώθηκε η αναθεώρηση του κανονισμού. Αυτό είναι αναγνώριση κάποιων ε, επεισοδίων, ε, κάποιων καταστάσεων όπου οι εταιρείε ε, αντιμετώπισαν απεριόριστες υποχρεώσεις αποζημίωσης στην ουσία. Όταν είναι δική μας ευθύνη, η πετιότητα, αποδεχόμεστα ότι θα πρέπει να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις. Αλλά σε ορισμένε περιπτώσεις πρέπει να φροντίσουμε για τους επιβάτες παρά το ότι η ευθύνη είναι αλλού γιατί δεν μας παρασχέθηκαν και μας υπηρεσίες για τις οποίες είχαμε συμβατική ε, σύμβαση. Θέλουμε να φροντίσουμε τους ε, επιβάτες, αλλά θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να μας επιστραφεί το κόστος αυτής της φροντίδας από τους πραγματικούς επαιτίους. Εάν θεωρήσουν ότι είναι άδικη αυτή η επιστροφή, τότε μπορεί να στραφούν εναντίον μας. Αλλά αυτό ε, αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης από τον ε, αερομεταφορέα που πληρώνει τον καταναλωτή στο τρίτο μέρος. Και ήδη έχουν δυνατότητα να στραφούν εναντίον μας. Όπως βλέπετε οι, οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας μπορούν να στραφούν εναντίον μας και τα αεροδρόμια μπορούν να στραφούν εναντίον μας εάν θεωρήσουν ότι τελικά ε, υπέστησαν μεγαλύτερο κόστος. Υπάρχει λοιπόν κάποια ανάγκη εξισορρόπησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τις εταιρείες charter και τους ε, ε, οργανισμούς ε, οργανωμένων ταξιδίων. Παρακαλώ, ο κύριος Μπάουλ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συμβάλλουμε. Η εταιρεία του, η Travel PLC, είναι μία από τις μεγαλύτερες, ε, τους μεγαλύτερους ομίλους ε, ταξιδιών αναψυχής. Ε, έχουμε ε, κεφάλαια γύρω στα 40 δις, 54.000 εργαζόμενους, κυρίως στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ε, ε, σοβαρή δέσμευση και σοβαρή συμβολή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Να μερικέ από τι εταιρείε μα. Βλέπετε εδώ το χαμόγελο που είναι το λογότυπό μα. Όπου υπάρχει αυτό το χαμόγελο είναι TUI. Και να μερικέ από τι εταιρείε ε, που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μα. Εμεί πηγαίνουμε του Ευρωπαίου από το κρύο της Βόρειας Ευρώπης στη Νότια Ευρώπη και ακόμη μακρύτερα. Έχουμε τη δική μας αεροπορική εταιρεία. Αλλά ε, το γονιδιωμά μας είναι πάροχος οργανωμένων ταξιδίων, οργανωμένων διακοπών. Πολλές πωλήσει γίνονται μέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω ε, ε, γραφείων που έχουμε και άλλων ταξιδιωτικών πρακτόρων. Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις τώρα. Δυστυχώς δεν είναι οι, οι, εταιρείε όλες ε, ίδιου τύπου. Οι εταιρείε charter χρειάζεται να πληρώσουν περισσότερες αποζημιώσεις αναλογικά. Ζητήσαμε από την KPMG μία ε, ανεξάρτητη μελέτη που κοίταξε πώς τα διάφορα τμήματα των αερομεταφορέων ε, ε, υφίστανται τι καθυστερήσει 2011 2011-2012. Βλέπετε εδώ πως δεν είναι μικρή διαφορά. Βλέπετε ότι ο τομέα charter, ναυλωμένων πτήσεων, ε, έχει τρει με τέσσερι φορέ παραπάνω καθυστερήσει από του άλλου αερομεταφορεί. Γιατί άραγε, για δύο λόγου. Περισσότερε καθυστερήσει έχουν οι πτήσει charter, γιατί εμεί δεν ακυρώνουμε πτήσει. Γιατί δεν τι ακυρώνουμε. Έχουμε υποχρέωση προ του πελάτε. Με βάση το οργανωμένο ταξίδι και την οδηγία που τα καλύπτει, πηγαίνουμε προ ε, ε, ε προορισμού που έχουν λιγότερη πυκνότητα πτήσεων και με μεγάλη πληρότητα. Εάν λοιπόν ε, δεν γίνει μια πτήση όπως πρέπει, δεν μπορούν να την ακυρώσουν. Γιατί οι πελάτες του δεν έχουν στην πράξη καμία δυνατότητα αλλαγή δρομολογίου. Τι σημαίνει αυτό? οποιαδήποτε διακοπή πτήσεων δεν είναι μία μόνο ακύρωση, είναι μια σειρά από, μακρο, μακριού μήκους καθυστερήσεις. Οι εταιρείε charter δεν μπορούν να αλλάξουν πολύ το πρόγραμμά τους. Πηγαίνουν, ε, ξεκινάνε από μικρά περιφερειακά αεροδρόμια προς μικρά άλλα αεροδρόμια, όπου οι δυνατότητες επισκευών, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο περιορισμένες. Αυτά είναι στοιχεία που οδηγούν σε περισσότερε καθυστερήσει, γιατί δεν υπάρχουν αρκετέ δυνατότητε να καλυφθούν οι καθυστερήσει και υπάρχουν λιγότερε δυνατότητε να αλλάξει κανεί, για παράδειγμα, αεροπλάνο για να καλύψει μια καθυστέρηση. Παράλληλα, οι επιβάτε μα καλύπτονται, προστατεύονται καλύτερα με βάση την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια και επειδή είναι ταξιδιώτε ανα, αναψυχής μπορούν να ανεχθούν περισσότερη καθυστέρηση από ότι οι επιβάτες που πηγαίνουν για δουλειά κάπου. Και επιπλέον οι εταιρείε μας ε, φροντίζουν καλύτερα τους ε, πελάτες, αν υπάρχει καθυστέρηση, ενημερώνουν τους πελάτες, αν η πτήση επιστροφής ε, καθυστερήσει, θα υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω μεταφοράς. Τι λύση υπάρχει λοιπόν, δύο δυνατότητες. Ή θα εξαιρεθούν από τον κανονισμό 261 και θα μείνουμε στην οδηγία ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε το καθεστώς που θα εφαρμοστεί να ε, είναι λελογισμένο όσον αφορά τις ε, αποζημιώσεις. Εάν είναι δυσανάλογο το καθεστώς θα έχει τρομερά ε, απροσδόκητες ε, επιπτώσεις. Εμείς πηγαίνουμε σε μικρότερα δρόμια, υποστηρίζουμε τον τουρισμό στις περιφερειακές οικονομίες και δίνουμε περισσότερη προστασία στους πελάτες. Εάν είναι δυσανάλογο το καθεστώς αποζημιώσεων, θα απειληθούν όλες αυτές τις δυνατότητες. Ανάλογες πρέπει να είναι τώρα κυρίως ως προς τι. Ανάλογες με το κόστος ε, του ταξιδίου. Εδώ βλέπετε η μέση τιμή μας για τα διάφορα είδη πτήσεων. Ας πάρουμε τη μέση περίπτωση μέσης διάρκειας της 861 ευρώ. Καθυστέρηση, αποζημίωση για καθυστέρηση 400, ποσοστό 46%. Εάν έχετε καθυστέρηση και ε, όταν ε, ε, πάτε στην, στον τόπο διακοπών και όταν επιστρέφετε, στην ουσία έχετε πάρει αποζημίωση το κόστος των διακοπών σας. Αυτά είναι τα κυρία σημεία. Τα σημεία ενεργοποίησης για τις αποζημιώσεις 5, 9 και 12, λογικό αλλά ε, οι διάφορες λωρίδες ε, αποζημίωσης πρέπει να ε, σχετίζονται με αυτά τα κατόφλια ενεργοποίησης. Και επίσης πρέπει οι έκτακτες περιστάσεις να έχουν να κάνουν με τις τοπικές συνθήκες. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην πλευρά των καταναλωτών. Έχουμε ε, δύο ομιλητές. Πρώτον από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών, Γιολάντα Γκέρζλ, που διευθύνει το σουηδικό γραφείο του δικτύου. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών που μας κάλεσε ε, να μιλήσουμε για την άποψη των καταναλωτών. Ε, ε, έχουμε μια σύντομη παρουσίωση του δικτύου κέντρων καταναλωτών. Το δίκτυο έχει 28 κρατημέλη. Η Κροατία ε, θα προσχωρήσει τον 1η Ιουλίου 2013 και θα έχουμε και την Νορβηγία και την Ισλανδία. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Έχουμε, ασχολούμεθα με τις μεταφορές τις διασυνοριακές. Παρέχουμε Πληροφορίε πληροφορίες και συμβουλές για τα δικαιώματα των καταναλωτών και επίσης βοήθεια για την διεκπαιρέωση των διασυνοριακών καταγγελιών και προωθούμε επίσης την, επίλυση την αλλακτική επίλυση διαφορών. Έχουμε εκστρατείες δημόσιες πληροφοριών, έρευνες, δημοσιεύσεις, διαβουλεύσεις. Το 2012 είχαμε 72.067 επαφές, 32.107 ήταν καταγγελίες και και 32% αφορούσαν τον τομέα των μεταφορών, από τις οποίες 21,6 επιβάτες αεροπορικών γραμμών. Ε, πώς ε, μοιραζόμαστε τις καταγγελίες, ερχόμαστε σε επαφή με τον καταναλωτή, επίσης ε, και τον μεταφορέα. Ποιος έχει την άμεση επαφή με τον αερομεταφορέα στην ενδιαφερόμενη χώρα αν όλα πάνε καλά, επιλύονται οι ε, περιπτώσεις, αλλά αν τα πράγματα στραβώσουν, ε, ε, θα έχουμε μια εναλλακτική επίλυση διαφορών αυτό το σύστημα και επίσης τα όργανα επιβολής, τα εθνικά και έχουμε επίσης μια, μια συνεργασία προστασίας καταναλωτών. Εμείς είμαστε στη Σφυδία το εθνικό όργανο επιβολής βεβαίως είναι οι απόψεις μας. Έχουμε δυσκολίες στο, στη διεκπαιρέωση των καταγγελιών, στην επίλυση των διαφορών λόγω των διαφορών στην ερμηνεία του νομοθετήματος. Επίσης, το πρόγραμμα της αλλαγής δρομολογίου και η επιστροφή σε περίπτωση ματαιωμένων πτήσεων εξαρτάται από την καλή θέληση των εταιριών. Η βοήθεια, η αρρωγή, η ανισότητα στην μεταχείριση, έλλειψη πληροφοριών, οι απατηλές πληροφορίες στους καταναλωτές αναφέρονται. Έχουμε προβλήματα με την αφαιρεγγιότητα, με την πτώχευση των αεροπορικών εταιριών. Είχαμε πολλές περιπτώσεις πέρσι, έχουμε διάφορες λύσεις, είναι ένα κρίσιμο θέμα σχετικά με τα δικαιώματα των επαγωτών. Έχουμε τις καθυστερήσεις πτήσεων. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα είναι η άρνηση των αερομεταφορέων να ε, αναγνωρίσουν ε, την περίπτωση Sturgeon ε, και έχουμε δυσκολίες για την ερμηνεία, την εκτίμηση ε, των εκτάκτων περιστάσεων και αναφέρομαι στην υπόθεση Valentine δεχόμαστε την πρόταση αναθεώρησης, τροποποίησης του κανονισμού. Έχουμε μερικά θέματα. Πιστεύω, ξέρουμε ότι ο κανονισμός δεν ισχύει για τους ίδιους κανόνες καταγγελιών όπως η Σύμβαση Μόντραν άρθρο 47, αλλά ε, οι απαιτήσει μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα μέρη. Έχουμε εναρμόνιση. Η εναρμόνιση των κανονισμών θα είναι ωφέλιμη για όλους. Επίσης, ε, η Νομίζω ότι ε, οι πτήσει ε, θα μπορούσαν ε, να περιληφθούν οι πτήσεις, οι περαιτέρω πτήσεις θα μπορούσαν να περιληφθούν στη νέο 261 επειδή υπάρχουν προβλήματα των καταναλωτών όπως για την αραγή, αρρωγή στο άρθρο 66. Η προθεσμία για τις καταγγελίες θα πρέπει να μετρά από το μόλις ο επιβάτης δεχθεί τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα δικαιώματά του. Είναι, είναι καλό να έχουμε ε, διευκρινισμένη την αντίληψη των εκτάκτων περιστάσεων στο παράρτημα 1 του κανονισμού, αλλά πιστεύουμε ότι παραδείγματα στο παράρτημα είναι πολύ γενικά και δεν είναι σαφή ως προς τι είναι οι έκτακτες περιστάσεις. Όταν λοιπόν μια περίπτωση εμπίπτει στην κατηγορία των εκτάκτων περιστάσεων πρέπει να βασίζεται σε ορισμένους όρους. Ε, νομίζουμε ότι η προθεσμία των τριών ωρών είναι λογική ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναθεώρηση να βασίζεται στην υπόθεση Sturgeon. Ξέρω και η οργάνωσή μας αναγνωρίζει βεβαίως ότι οι αποζημιώσεις είναι οικονομική επιβάρυνση για τους αερομεταφορείς, αλλά θα πρέπει να υπερέχουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα άλλα θέματα προς εξέταση, η διευκρίνηση ότι οι αερομεταφορείς δεν μπορούν να περιορίσουν την αλλαγή δρομολογίου στη δική τους εταιρεία, θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 8 ε, τι σημαίνει η αλλαγή δρομολογίου χρησιμοποιώντας άλλα μέσα. Ποιες, νομίζουμε ότι η έκφραση συγκρίσιμη όρη μεταφοράς ε, είναι κάτι το ασαφές. Νομίζουμε ότι 12 ώρες το όριο είναι πάρα πολύ μακρύ. Θα πρέπει η περίοδος ακυρώσεως να συνδέεται με την διάρκεια της πτήσης ούτως ώστε να αντανακλά ε, την ζημία που επιβαρύνει τον επιβάτη πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες δεσμευτικές, ούτως ώστε να παρέχονται πληροφορίες ε, είτε ο επιβάτης περιλαμβάνεται σε μία συμφωνία ή σε πολλές συμφωνίες και να λαμβάνεται υπόψη επίπτωση πάνω στα δικαιώματα των επιβατών. Επίσης, ε, ο ορισμός της νύκτας ε, πρέπει να αρχίζει στις 10 ε, η ώρα το βράδυ, ότι πάρα πολλοί επιβάτες χρειάζονται ξενοδοχεία πριν από τη 12η, από τα μεσάνυχτα. Βεβαίως οι απαιτήσει για προγράμματα έκτασης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μικρότερα αερολιμένες ο περιορισμός σε μεγάλα αεροδρόμια δεν λαμβάνει υπόψη τις, τα συμφέροντα των καταναλωτών. Έχουμε εμεί στη Σουηδία τον Κότεμπορ και μικρά αεροδρόμια που δεν πληρούν τα κριτήρια. Άρθρο 7 νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια προσθήκη ότι ο επιβάτης θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο της πληρωμής διότι πολύ συχνά πληρώνονται με επιταγές, με ένα βάουτσερ και ε, συνδέεται με ένα κόστος ε, και τότε δεν λαμβάνουν αποζημίωση οι επιβάτες. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να επιτρέπει στις εταιρείε ε, να παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις συνάπτοντας εθελοντικές συμφωνίες με τον επιβάτη. Συστηματικά την χάνουν εκμετάλλευση οι επιβάτες, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι όροι και τα δικαιώματα των επιβατών βάσει του κανονισμού. Είναι, θα πρέπει τα δικαιώματα να τηρούνται. Άρθρο 9, σημείο 4. Η προτινόμενη περιορισμό των τριών νυχτών είναι κάτι το λογικό προς το συνολικό κόστος του καταλήματο. Νομίζω ότι το ποσό θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τιμές των ξενοδοχείων που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο. Αυτό εξαρτάται από την χώρα. Άρθρο 11, 3 ε, τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ε, θα πρέπει να αναφέρουν οποιοδήποτε ειδική ανάγκη πριν από την ώρα αναχώρησης. Πιστεύουμε ότι Έχουμε τον κανονισμό 1107 του 2006 που αναφέρει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες δεν αναφέρουν ότι χρειάζονται βοήθεια 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Θα πρέπει να καταβληθούν ε, προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχει όμως τέτοια πρόβλεψη. Στο άρθρο 1 ο ορισμός των, των ατόμων με ειδικέ ανάγκε, ατόμων με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα, ο ορισμό αυτό δεν διευκρινίζεται. Θα πρέπει και στο άρθρο 5 τα σχέδια έκτακτη ανάγκη θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά σε άτομα με αναπηρίε και περιορισμένη κινητικότητα. Άρθρο 14.3 η υποχρέωση ενημέρωση των επιβατών σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι περιορισμένη σε άτομα τα οποία είναι σε τυφλά άτομα ή που δεν βλέπονται καλά, θα πρέπει όλα τα άτομα να ενημέρονται. Άρθρο 14, ο, ε, ο οργανισμός του αερολιμένα θα πρέπει να είναι υπεύθυνο ε, για τις ε, πληροφορίες στο αεροδρόμιο σχετικά με την άρνηση επιβίβασης. Θα πρέπει να υπάρχει κοινή ευθύνη με όλους τους άλλους φορείς. Άρθρο 16 θα πρέπει απαιτήσει ενημέρωση για τους αερομεταφερεί να περιλαμβάνουν τους μεσολαβητές των προγραμματισμένων ε, πτήσεων και των ομαδικών ταξιδίων. Δεν είναι μόνο ο αερομεταφορέας ε, της πτήση όπως στο άρθρο 45 της Σύμβασης του Μοντρεάλ ε, πάρα πολλοί αερομεταφορείς ε, νοικιάζουν ε, άλλες αερογραμμές και αεροπλάνα για, ε, για πτήσεις και έχουν κοινέ συμφωνίες με άλλους μεταφορείς. Δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο όταν υπάρχουν προβλήματα. Επίσης, ο χρόνος, η προθεσμία των τριών μήνων στο άρθρο 16α σημείο 2 ε, δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μπορεί για διάφορους λόγους ο επιβάτης δεν μπορεί μέσα στην προθεσμία αυτή ε, να αξιώσει ε, μια αποζημίωση. Μπορεί εξάλλου να μην έχει ενημερωθεί μόλις Μόνο θα πρέπει η προθεσμία να αρχίσει να τρέχει όταν ο επιβάτης έλαβε τις πληροφορίες για τα δικαιώματα του. Μπορείτε να κλείσετε, λέει ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι δωρεάν η καταγγελία για τους επιβάτες και να έρχονται σε επαφή με τους αερομεταφερείς και θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διάφοροι όροι σχετικά με τις καθυστερήσεις. Τελευταία διαφάνεια, το θέμα ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ταξιδεύουν με ασφάλεια γνωρίζοντας ότι οι εταιρείε θα τηρούν τα δικαιώματά τους και ότι οι κανόνες θα ισχύουν εξίσου για όλες τις αεροπορικές εταιρείε Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο σας. Γι' αυτό κλείνω. Ευχαριστώ. Next from the European... Επόμενη ομιλήτρια η Ούρσουλα Πάχλ, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών, BEUC. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ την Επιτροπή που κάλεσε ε, τη δική μας οργάνωση σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, λέει η ομιλήτρια. Είμαστε ένας οργανισμός ε, που αποτελείται από 41 εθνικές οργανώσεις καταναλωτών. Οι αερομεταφορείς υπογραμμίζουν ότι έχουν πολύ συνεκτική θέση και εμείς το ίδιο και σας διαβεβαιώ ότι είναι ενωμένη η θέση μας ως προς τη θέση ως προς τις 41 οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών τις οποίες εκπροσωπούμε εδώ σήμερα. Πριν ξεκινήσω ε, το σχολιασμό για τα διάφορα ζητήματα, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, μια γενικότερη παρατήρηση, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την αναθεώρηση. Πολύ συχνά από πλευράς καταναλωτών λέγεται κάτι που είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Έχουμε όλο και περισσότερες καταγγελίες, όλο και περισσότερα παράπονα στις εναρίες μεταφορές. Υπάρχουν προβλήματα με την ερμηνεία των κανόνων. Συστηματικά αναθεωρείται η δυνατότητα των αερομεταφορέων να προσφέρουν τη φροντίδα, τη στήριξη και την αποζημίωση που οφείλουν στους καταναλωτές. Ο αριθμός των καταγγελιών έχει αυξηθεί κατά 96% τα τελευταία πέντε χρόνια. Εντυπωσιακά είναι και τα αριθμητικά στοιχεία που μας δίνουν τα δικά μας μέλη. Το μέλος μας από το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε μια έρευνα το 2010 η οποία έδειξε ότι το 44% των επιβατών με σημαντικές καθυστερήσεις δεν έλαβε καμία φροντίδα, καμία βοήθεια. Το μέλος μας από τη Δανία μας είπε ότι μόνο το 4% των επιβατών που καθυστέρησαν έλαβαν τελικά αποζημίωση για τις καθυστερήσεις μόνο το 2% ε, ε, έλαβε αποσμίωση για την ακύρωση και αντίστοιχα στοιχεία έχουμε από το μέλος μας από την Γερμανία και μόνο εάν ο επιβάτης το ζητούσε αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα, ποιο είναι το σημαντικό για τον επιβάτη. Να έχει την εμπιστοσύνη ότι ο αερομεταφορέας θα σεβαστεί τη συμφωνία ώστε να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του εγκαίρος και ότι αν προκύψουν προβλήματα, εάν υπάρξει καθυστέρηση ή διακοπή του ταξιδιού, να νιώθει εμπιστοσύνη ότι κάποιος θα τον φροντίσει. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το οποίο θα πετύχουμε με την αναθεώρηση έτσι όπως διατυπώνεται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, ισχυρές είναι οι ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν ε, στο γεγονός ότι εάν περάσει η αναθεώρηση θα αποδυναμώσει δικαιώματα που έχουν ήδη κατοχυρωθεί και παγιωθεί και προβλεφθεί μάλιστα και από το δικαστήριο. Η μη συμμόρφωση από πλευράς κλάδου θα επανέλθει διότι θα μειωθούν οι υποχρεώσεις τους και η αξιολόγηση αντικτύπου ε, δείχνει μάλλον ότι οι λιγότερες υποχρεώσεις θα αποδυναμώσουν και το κίνητρο για συμμόρφωση. Ε, δεν είναι η σωστή βάση για να προχωρήσουμε κατά τη δική μας άποψη. Ποια είναι τα βασικά δικαιώματα τα οποία τίθενται ένα αμφιβόλο. Ε, το δικαίωμα στην αποζημίωση για μεγάλες καθυστερήσεις Καταρχήν είναι καλό αυτό, αλλά έχει διασπαστεί σε τρία κατόφλια εξαιρετικά μεγάλα, στις 5 ώρες, στις 9 και στις 12 ώρες, ε, αντιβαίνοντας την απόφαση ε, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Δικαστηρίου που προβλέπει αποσημείωση μετά τις 3 ώρες. Ε, καθυστέρησης. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλό αυτό, πιο ευνόητο, πιο εύληπτο και για τους καταναλωτές και είναι και πιο εύκολο για τους αερομεταφορείς να το εφαρμόζουν. Δηλαδή υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης μετά από καθυστέρηση τριών ωρών. Δεν είναι πιθανή η εξήγηση της Κομισιόν ότι αν διατηρηθεί το τρίωρο αυτό θα υπάρξουν περισσότερα προβλήματα και θα ακυρωθούν περισσότερες πτήσεις. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Από εκεί και πέρα το δικαίωμα ε, για βοήθεια σε ε, εξαιρετικές συνθήκες η μείωση, η αποδυνάμωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων στα 100 ευρώ ανανύχτα και στις τρεις νύχτες διαμονή τριών ε, νυχτών θα φέρει τους επιβάτες σε δύσκολη θέση δεν είναι αναλογική αυτή η απάντηση στις εξαιρετικές περιπτώσεις που, και συνθήκες που δημιουργήθηκαν, για παράδειγμα με τον έφος ηφαιστειακής ε, τέφρας. Θεωρούμε ότι οι καταναλωτές θα δυσκολευτούν εξαιρετικά ε, να βρουν δωμάτιο ξενοδοχείου με 100 ευρώ τη, βραδιά ε, σε χώρες που δεν γνωρίζουν, που, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, χωρίς να ξέρουν τις τιμές της τοπικής αγοράς, θα πάρουν ό,τι τους προσφερθεί εκεί όπου έχουν ξεμείνει και τελικά θα καταλήξουμε να έχουμε επιβάτες να ε, διανυκτερεύσουν στο δρόμο λόγω αυτού του προβλήματος. Ως προς το την αλλαγή δρομολογίου, ε, καταρχάς είναι θετικό το ότι το συμπεριέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, 12 ώρες αναμονή πριν να συμμετάσχει στην αλλαγή δρομολογίου είναι με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα όταν βρίσκεται κανείς σε ένα σημείο που δεν έχει και πολλές αναχωρήσεις πτήσεων ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να προσφέρεται αυτή η ευκαιρία στον νωρίτερα αποφεύγοντας και την υποχρέωση ε, παροχής στέγασης αλλά θα πρέπει να είναι και επιλογή για τις μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι ο μόνος τρόπος ο επιβάτης να φτάσει στον προορισμό του τελικά ε, το συντομότερο δυνατό. Τώρα ως προς την πολιτική no show, όταν δεν εμφανίζεται ο επιβάτης ε, στη πτήση, έτσι όπως ε, είπε ο ε, πρόσωπος της ΙΑΤΑ. Διαφωνώ καθέτος, δεν είναι ψευδές το δικαίωμα αυτό του επιβάτη. Έχουμε διαφορά στην ερμηνεία. Υπάρχει μια σειρά δικαστικών αποφάσεων οι οποίες ξεκάθαρα προβλέπουν ότι η πολιτική non-show σύμφωνα με την οποία ο επιβάτης ε, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο για ένα σκέλος ενός εισιτηρίου ολόκληρου που έχει ήδη αγοράσει στο σύνολό του από πριν είναι αθέμητη πρακτική και δεν μπορεί να ε, ε, υπάρχει να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε σύμβαση για την αγορά και πώληση καταναλωτικού προϊόντος. Εμείς θέλουμε να απαγορευτεί πλήρως η χρήση της ρήτρα no-show στις συμβάσεις που συνάπτουν οι εταιρείε με τους καταναλωτές από εκεί και πέρα, οι εξαιρετικέ περιστάσεις, συμφωνούμε, είναι πολύ δύσκολο και περίπλοκο αυτό το θέμα. Ε, καλωσορίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση όμως που υποβάλλει ε, δίνει λαβή για ακόμα πιο πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Και ο κατάλογος των ε, κατεξαίρεση συνθήκων και περιστάσεων είναι εξαιρετικά εξαντλητικός. ο οραματοφορέας οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε εύλογη προσπάθεια να αποφύγει την ε, ε, ταλαιπωρία ή το πρόβλημα εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στο κείμενο. Σίγουρα η πρόταση της Κομισιόν έχει και θετικά στοιχεία. Καλύπτονται οι πτήσεις ανταπόκρισης τις οποίες δεν προλαβαίνουν οι επιβάτες. Υπάρχει το rerouting, η αλλαγή δρομολογίου. Μπορεί κανείς να διορθώσει τυπογραφικά, ορθο, ορθογραφικά λάθη στο όνομά του χωρίς να πληρώσει και είναι απαραίτητο το να εφαρμόζονται όλα αυτά με πιο αποτελεσματικό τρόπο να υπάρξει περισσότερη πρόβλεψη για νομοθετική ως προς τις καταγγελίες των καταναλωτών. Αυτή η διάρκεια, η προθεσμία των ε, τριών μηνών ε, ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμεραγκ εις βάρος των καταναλωτών. Και δύο στοιχεία που θέλω να αναφέρω είναι τα εξής. Η πολιτική no-show είναι η κορυφή του παγόβουνου ως προς την αθέμητη καταναλωτική και εμπορική πρακτική. Έχει γίνει πολύ εντατική δουλειά και δαπανηρή. Άνθρωποι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές εναντίον ε, εταιριών με βάση τις συστάσεις της ΙΑΤΑ και έχουμε διάφορες δικαστικές αποφάσεις σε διάφορα κράτη-μέλη που έχουν ήδη εκδοθεί και ειδικής ενδεχομένω. Ε, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αυτή τη μαύρη λίστα. Να ε, συνεχίσετε να υποβάλλετε αυτό το αίτημα γιατί είναι σημαντικό και ως προς την αφαιρεκιότητα όπως είπε και η Γιολάντα κάτι το σημαντικό για τους καταναλωτές. Δεν είμαστε καθόλου πεπισμένοι ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν η πρόσφατη για τα εθελούσια μέτρα που λαμβάνονται ότι αρκεί αυτό. Θα θέλαμε να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας ε, ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρεία θα προβλέπεται ο επαναπατρισμός και τα διάφορα τα υπόλοιπα. Είναι γεγονός ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη και είναι αρκετές. Είναι τρομερό αυτό ότι ε, προτείνεται μια νομοθεσία η οποία δεν σέβεται ήδη υπάρχουσα νομολογία σε γενικές γραμμές δεν πρέπει να αποδυναμωθούν τα δικαιώματα των επιβατών και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει το παν για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις έτσι όπως τις περιγράψαμε στην παρέμβασή μας. Ευχαριστώ. Τα τώρα. Πρώτα απ' όλα οι σκιώδεις κυρία Βανόρ, η κυρία Σάβη και Για τον κύριο Τέιλορ, η κυρία Φώστερ. Όποιοι άλλοι συνάδελφοι παρακαλώ να το δηλώσουν. Μπένιον, μάλιστα. Εντάξει. Η κυρία Ζαναλόβα. Άλλος. Μπένιον και Ζανάλογα. Και οι τέσσερις σκιώδεις σύγητες. Η κυρία Βανόν. τέσσερα λεπτά. Η Μπερναντέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Βερνιό, λοιπόν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αναθεώρηση του κανονισμού και πολύ λεπτό το θέμα αυτό στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Διότι επειδή είμαι αρμόδια από πλευρά σοσιαλιστών και δημοκρατών για την προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, στην Επιτροπή Μεταφορών, για μένα πρέπει να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Αλλά παράλληλα να λάβουμε υπόψη και την πραγματικότητα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε. Οι εταιρείε, τα αεροδρόμια, να βρούνε ένα μόντους βιβέντη, ούτω ώστε ε, να συνεργάζονται για να βελτιωθεί η ενημέρωση και να εφαρμόζονται καλύτερα τα δικαιώματα των επιβατών χωρίς να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητες οικονομικές δυσχέρειες. Αυτό που διαπιστώνουμε και ως και το βλέπω, είδαμε ότι οι διάφοροι ενεχόμενοι του κλάδου με τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, τα αεροδρόμια, οι εταιρείε, τα αργωμένα ταξίδια και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, οι οποίοι καταναλωτέ δεν ενημερώνονται πολύ συχνά σωστά. Βεβαίω να υπάρχει, εάν υπάρξει ε, μεγάλη έκταση επεισόδιο, ένα ε, σχέδιο έκτακτη ανάγκη, πολύ καλή ιδέα. Αλλά Μεγάλο ερώτημα για το οποίο δικαίως πιστεύω ανησυχούν ε, τα αεροδρόμια. Ε, μήπως οι αεροπορικές εταιρείε ε, τους αναθέσουν τις δικές τους ευθύνες. Για παράδειγμα ότι τα αεροδρόμια θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαφή με τους επιβάτες. Και εάν για παράδειγμα δεν έχει κανείς τη δυνατότητα ε, να ε, επιβιβαστεί στην πτήση ε, επιστροφής αν δεν πάει στην πτήση μετάβασης. Εδώ υπάρχουν αντιθέμενες απόψεις και η τελευταία παρέμβαση, παρέμβαση της οργάνωσης καταναλωτών πρέπει μια για πάντα να προσαρμόσουμε τις καθυστερήσεις. Όλοι το είπαν, από όλες τις πλευρές. 12 ώρες 12 ώρες. Είναι υπερβολικό χρονικό διάστημα. Αν είναι κάποιος επιβάτης με την οικογένειά του, ε, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κατάλογο. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν ορισμό κάπως πιο συγκεκριμένο για το τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν τα πάντα και τίποτα αυτοί οι ορισμοί. Και επίσης η επαφή, η επαφή, η πληροφόρηση. Περισσότεροι επιβάτες όταν αγοράζουν ένα εισιτήριο. Και αυτό είναι ευθύνη των αερομεταφορέων. Όταν προσφέρουν ένα εισιτήριο πρέπει να προσφέρουν όρους και συνθήκες κατανοητούς, να καταλαβαίνουν ποια είναι τα δικαιώματά τους επιβάτες αν υπάρξουν προβλήματα, αν υπάρξουν καθυστερήσεις. Για τις αποσκευές τους οι χαμηλού κόστους εταιρείε, εταιρείες, που κι εγώ τις παίρνω ορισμένε φορές. Οι επιβάτες δεν έχουν υπόψη τους, δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα στο αεροδρόμιο. Κάποιος το, κάποιος το ανέφερε. Πάω με την τσάντα μου, με την τσάντα μου με όλα μου τα χαρτιά μέσα. Αγοράζω ένα δώρο, ένα άρωμα να κάνω. Όχι. Είμαι υποχρεωμένη να το βάλω στην τσάντα μου. Και αν είναι κάτι που δεν χωράει στην τσάντα μου πρέπει να το αφήσω έξω απαράδεκτο και δεν το ξέρουν οι επιβάτες εκ των προτέρων. Για τις υπόλοιπες ε, αεροπορικές εταιρείες, για τις αποζημιώσεις, είδαμε τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των ε, εταιριών ε, χαμηλού κόστους και των κανονικών εταιριών. Πρέπει να βρούμε το σωστό μέσο όρο να μην πω σε λεπτομέρειες γιατί και εδώ υπάρχουν ε, πολλές λεπτομέρειες που είναι θεμελιώδεις. Πρέπει να βρούμε το σωστό μέσο όρο και ακόμη δεν έχουμε βρει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάλιζα, τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο δεν θα πω πολλά ευχαριστώ και τέτοια. Επί της ουσίας. Νομίζω Νομίζω ότι οι προτάσει τη Κομισιόν για ορισμένα θέματα γέρνουν από τη μια, για ορισμένα την άλλη. Αποζημίωση μόνο μετά από πέντε ώρες εντός της Ευρώπης λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πτήσεις στην Ευρώπη δύο-δύο μισή ώρες. Ανησυχητικό επίσης είναι ότι σε έκτακτες περιστάσεις Οι έκτακτες περιστάσεις, εάν υπάρξει μηχανική βλάβη, είναι μόνο αν είναι σε αυτήν ή την προηγούμενη πτήση. Αλλά ξέρετε, εάν είναι μια μικρή εταιρεία και έχει μια μηχανική βλάβη στην πρώτη του πτήση το αεροσκάφος, μπορεί να επηρεάσει τις επόμενες πέντε. Το ίδιο ισχύει για άλλες μικρές εταιρείες, η αλλαγή δρομολογίου εντός 12 ωρών. Πολύ συχνά ε, οι μικρές εταιρείες πετάνε μεταξύ αεροδρομίων όπου δεν υπάρχουν νυχτερινές πτήσεις. Επίσης, ένα πρόβλημα με την πρόταση της Επιτροπής είναι ο ορισμός της ακύρωσης. Τι είναι ακύρωση. Εάν ο πιλότος διαπιστώσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή ένας επιβάτης αρρωστήσει και δεν μπορεί να προσγειωθεί για παράδειγμα για κάποιο λόγο για κάποιο λόγο υπάρχει, μπορεί να υπάρξει θέμα ασφάλειας πρέπει να το δούμε mm. Ορισμένες ρυθμίσεις ε, είναι μεν πολύ φιλικές προς επιβάτες αλλά είναι δυσανάλογες είναι πολύ δύσκολο οι εταιρείες να έχουν ε, στρατηγική πώληση των εισιτηρίων τους με αυτές τις ρυθμίσεις. Οι εταιρείε χαμηλού κόστους ε, πολλές φορές δεν έχουν ε, πτήσεις για επιστροφή. Για τις πτήσεις charter τώρα. Οι πτήσεις charter. Θα πρέπει να εξαιρεθούν μήπως. Να το δούμε αυτό. Ή να μείνουν με τον κανονισμό 9-10. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις πολύ μεγάλων καθυστερήσεων σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει επίσης να δούμε πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς είναι η χειραποσκευή, ε, πόσο είναι το βάρος των αποσκευών που, μπορούν να πάρουμε, που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας στο αεροπλάνο εκτός από τη χειραποσκευή. Ακούσαμε για παράδειγμα για τις αγορές στα αεροδρόμια. Πρέπει να υπάρξει πιο συγκεκριμένη ρύθμιση. Οι ανταποκρίσεις τώρα. Το συζητήσαμε επί μακρόν. Πρέπει να υπάρξει η σωστή αναλογία μεταξύ συντόμων και ε, μεγάλων πτήσεων. Η ενημέρωση των επιβατών ε, εγκαίρως όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, ακυρώσεις είναι επίσης πρωταρχική σημασίας. Πρέπει να λαμβάνουν όλη την αναγκαία πληροφόρηση για τι αποσκευέ του, για παράδειγμα. Όλη αυτή πρέπει να χορηγείται. Ήδη πριν ε, να φτάσει στο αεροδρόμιο ο επιβάτης πρέπει να ξέρει τι δικαιώματα έχει, τι μπορεί να πάρει στο αεροσκάφο κτλ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Θα ήταν πολύ καλό ε, όλοι μαζί να συνεργαστούμε ώστε ο κανονισμός ε, να έχει καλή κατάληξη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίχτενμπέργα, τέσσερα λεπτά. Κοιτάξτε, όταν ακούω αυτή τη συζήτηση, εδώ δεν μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά τα δικαιώματα των εταιριών έναντι των επιβατών, που πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ και όχι αντιστρόφως, ενώ αυτό υποτίθεται ότι επιδιώκαμε. Και είναι ήδη πολύ κακή η πρόταση της Επιτροπής και όταν ακούω και τις προτάσεις των εταιριών, τότε στο τέλος θα τα κάνουμε μουσκεμά. Μίλησα με δικηγόρους οι οποίοι μου λένε ότι 80% όλων των ε, παραπώνων που κάνουν οι επιβάτες δεν δικαιώνονται. Με τον νέο κανονισμό θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, οι επιβάτες πολλές φορές ε, δεν ε, μπορούν να πάρουν την πτήση τους και θεωρούνται και ενοχλητικοί επί από πάνω, αντί να θεωρούνται άτομα που πρέπει να βοηθηθούν. Με απογοητεύει ιδιαίτερα ότι τα άτομα μειωμένη κινητικότητα, για παράδειγμα, δεν βλέπω να βελτιώνεται καθόλου η κατάστασή του. Και είναι απολύτω επίγον και αναγκαίο. Έχουμε καταστάσει όπου οι αεροπορικές εταιρείε απαιτούν να τους στείλουν εκ των προτέρων ιατρικά πιστοποιητικά ότι είναι ανάπηροι. Εδώ πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Και ελπίζω η Επιτροπή μας να συμβάλλει για την έγκαιρη ενημέρωση. Την τελευταία φορά που καθυστέρησε μία πτήση μου. Ενημερώθηκα. Για πρώτη φορά έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου μισή ώρα μετά την, καθυστέρηση, την έναξη καθυστέρησης. Ενώ ήμουν ήδη στο αεροδρόμιο. Πολύ με βοήθησε να μάθω ότι έχει καθυστερήσει η πτήση. Ε, έκτακτες περιστάσεις δεν καθορίζονται καλύτερα. Ε, ανωτέρα βία δεν καθορίζεται. Ούτε τι σημαίνει τεχνική βλάβη. Όλα αυτά ε, αξιοποιούνται κάθε φορά για να μην δοθούν αποζημιώσεις. Κάτι ακόμη προσωπικό. Με εκνευρίζει ιδιαίτερα ότι κατηγορούνται περίπου οι επιβάτες ότι θελημένα προσπαθούν να λάβουν αποζημιώσεις λες και είναι εγκληματίες όταν προσπαθούν να ε, απαιτήσουν τα δικαιώματά τους. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Ο ένας επιβάτης ε, ε, ιδίως ε, όσοι χρειάζεται να πετάνε συχνά, στην ουσία είναι έρμεα των περιστάσεων. Δεν έχουμε καμία επιλογή. Αυτό είναι το αποφασιστικό. 15 φορές για παράδειγμα δεν έλαβα ούτε καν απαντήσεις στα ερωτήματα που είχα θέσει γραπτός και σταμάτησα να ρωτάω. Κοιτάξτε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν, να αυξηθούν τα δικαιώματα από τρει ώρε σε πέντε να πάει καθυστέρηση. Η ανωτέρα βία να καθορίζεται ασαφώ και όλε αυτέ οι γκρίζε ζώνε να ερμηνεύονται στην ουσία κατά των επιβατών. Είναι πολύ λυπηρά όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν ε, βλέπουμε ότι 80% των περιπτώσεων όπου ζητείται αποζημίωση δεν δικαιώνονται, δεν καταλαβαίνω πλέον διότι ξέρετε δεν είναι αυτός σκοπός οι αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχει για να μετακινούνται οι επιβάτε. Με συγχωρείτε που τα λέω έτσι έξω από τα δόντια, αλλά αυτά που άκουσα σήμερα από τους εκπροσώπους του κλάδου ήταν λυπηρές. Ένας δικαστής δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει εάν ε, ε, έχει ε, δικαίωμα λόγω του επίπεδου των συζητημάτων του ένας πελάτης αποσμίωση, δηλαδή θα πρέπει να υποβάλει και τη φορολογική του δήλωση για να αποδειχθεί ότι έχει έννοια να πάρει κάποιο ποσό για αποσμίωση. Είναι πολύ προβληματικά όλα αυτά. Και κάνω έκκληση, κάνω έκκληση και καταλήγω, κάνω έκκληση. Έχετε στην ουσία σε τελευταία ανάλυση μονοπωλιακή δομή στην Ευρώπη. Εάν παρόλα αυτά Θέλετε επιπλέον να υποβάλλετε τους επιβάτες σε περαιτέρω ταλαιπωρία, τότε πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να πάω και σε μια άλλη επιτροπή όπου πρέπει να παρουσιάσω ένα θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Φώστα, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω όλοι θα μπορούσαμε ε, να πάμε σπίτι μας ε, να αφήσουμε εφόσον δεν θα έχουμε κανέναν που θα λειτουργεί τα περιφερειακά ε, αεροδρόμια. Ε, λυπούμε κυρία Γκέρσελ. Έχω εργαστεί ε, για την περισσότερο χρόνο της ζωής μου σε αυτόν τον κλάδο και είδα πόσο μεταχειρίζονται τους επιβάτες. Δεν πρέπει να συγχυστεί αυτό πρέπει να προσφέρετε μια, ένα καλό προϊόν, μια, μια καλή υπηρεσία στον καταναλωτή. Πώς, καν πώς αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που είναι εκτός κανόνα, πώς, αντιμετωπι, πώς αντιμετωπίζουμε έναν καταναλωτή σε ένα κατάστημα, σε ένα λεωφορείο. Έχουμε μια σύμβαση κατά κάποιο τρόπο, θα πρέπει να έχουν μια καλή συμφωνία περί αυτού πρόκειται και νομίζω ότι υπάρχει μια υποχρέωση και από τις δύο πλευρές να εξασφαλίσουμε ότι η σύμβαση αυτή, η συμφωνία αυτή τηρείται. Βεβαίως Υπάρχουν ορισμένα πράγματα ε, τα, και εναπόκειται στις, ε, στους αερολιμένες και στους αερομεταφορείς να δίνουμε τις καλές ε, πληροφορίες, να ασχολούνται με τις υπηρεσίες εδάφους, με τις αποσκευές. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ξέρει ο καταναλωτής ποια είναι τα προϊόντα σας, ποιες είναι οι υπηρεσίες σας, τι γίνεται με τις καθυστερήσεις. Βρίσκεται στα μισά του δρόμου. Ε, βεβαίως, ε, ε, ότι τι θα κάνουμε του χρόνου ερχόμενοι εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει ίσως να κολυμπάμε στην ε, μάχη αν δεν, δεν υπάρχει επιλογή διότι δεν έχει ε, μείνει τίποτα, εμείς θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν σημασία. Θα πρέπει έχουμε καλές εξυπηρετήσεις ε, και στις περιφερειές μας, όχι μόνο στους βασικούς κόμβους τους αεροπορικούς. Αυτό ε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια τιμωρητική στάση. Όχι. Αυτές, αυτά είναι τα θέματα που με ανησυχούν. Θα πρέπει να βρούμε έναν πρακτικό τρόπο να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι οι συγητής ε, είχε μια καλή παρουσίαση. Η Επιτροπή ανέφερε μερικά καλά σημεία και εμείς ζητήσαμε ορισμένες ε, διευκρινήσεις. Βεβαίως από την πλευρά των αερομεταφορέων μας ε, δώσαν ορισμένα παραδείγματα. Το interlining, δεν θέλω να απειληθεί το interlining, αυτή η συνεργασία μεταξύ των γραμμών. Χρειαζόμαστε λοιπόν βεβαίως αυτή την βελτίωση στους αερομεταφορείς Βεβαίω, οι άνθρωποι ε, φτάνουν σε ένα αεροδρόμιο και μετά πρέπει να ξανακάνουν έτσι εκείνο όταν έχουν να πάρουν μια περαιτέρω πτήση. Και επίσης ε, δεν λαμβάνονται υπόψη επιπτώσεις νοκών. Ε, μπορεί βεβαίω να υπάρξει μια καθυστέρηση που να επιβαρύνει κατά μια μέρα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό. Σχετικά με τα charter τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν ακυρώνουν ε, διότι πηγαίνουν σε απομακρυσμένα σημεία και θα πρέπει να φροντίσουν τους επιβάτες διότι θα πρέπει να πάνε στον προορισμό τους να επιστρέψουν. Ε, δεν ξέρω ε, ότι θα πρέπει να έχουμε αυτά τα ομαδικά ταξίδια στον κανονισμό 261. Ε, θα πρέπει να δούμε τους διάφορους ε, ορισμούς βεβαίως. Βεβαίως, καμιά φορά όλες τα καθίσματα είναι άδεια. Βεβαίως έχουμε τις διευκρινήσεις για την αλλαγή του, της ορθογραφίας του ονόματος Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβετε εμπορικέ αποφάσει και υπάρχουν επίση και υποχρεώσεις από την πλευρά των καταναλωτών. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσε οι παρουσιάσει που κάνατε και οι διευθυνήσεις τη Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Αν ε, θέλετε να μείνετε στον κλάδο αυτό, στη δραστηριότητα αυτή, θα πρέπει να καταβάλλετε προσπάθειες και θα πρέπει η Επιτροπή να συνεργαστεί με τον εισηγητή ε, για να έχουν επιλογή οι καταναλωτές, για να μείνουν οι άνθρωποι στην ε, δουλειά τους και θα πρέπει να μπορούμε να ερχόμαστε εδώ από καιρού καιρών με ένα αεροσκάφος, κύριε Μπάνιαν. Δύο λεπτά. Μερικά σημεία θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι τα δικαιώματα είναι δίκαια, τα δικαιώματα τόσο των εταιριών όσο και των επιβατών, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν ε, σχετικά με το σύστημα αυτό, hub and spoke, ε, ενδιαφέρον, δεν δεν πρέπει βεβαίως να θέσουμε σε κίνδυνο ε, την κατάσταση. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία ανέφερα και εγώ. Βεβαίως είναι σωστό οι ε, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους να έχουν όρια ε, σχετικά με τις ε, χειραποσκευές, αλλά θα πρέπει να είμαστε επίσης και ορθολογιστικοί. Βεβαίως ε, ταξιδεύουμε όλοι πιο ελαφρά ε, και όλοι περισσότεροι αν θέλετε επιβαρυνόμαστε, τιμωρούμαστε έχοντας μία αποσκευή διότι κυρίως οι γυναίκες με τις μικρές τους τσάντες δεν μπορούν να βάλουν ε, πολλά πράγματα. Βεβαίως αν μπορεί κανείς να βάλει δύο τσάντες μέσα στην αποσκευή είναι καλύτερο. Σχετικά με την αλλαγή δρομολογίου και τι ανταποκρίσει, νομίζω ότι είδαμε πως χρησιμοποιώντας πολλά μέσα μπορεί κανείς να αλλάξει δρομολογείο. Βεβαίως μπορεί κανείς ανάμεσα στο αεροπλάνο και στο τρένο να έχει ε, τώρα ένα συνδυασμένο ε, εισιτήριο. Όταν φτάνει κανείς στο Charles de Gaulle τώρα, η Air France ε, του, δίνει ένα εισιτήριο σιδηροδρομικό για να φτάσει στο Στρασβούργο. Βεβαίως δεν ξέρω τι γίνεται με τα τρένα αν παίρνει κανείς αποζημίωση. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αλλαγή δρομολογίου που χρησιμοποιεί δύο ε, μέσα μεταφοράς. Τα άτομα ε, τα οποία πηγαίνουν, ταξιδεύουν ε, σε, για μια συνάντηση και επιστρέφουν την ίδια μέρα αν έχουν πέντε ώρες καθυστέρηση ματαιώνεται όλος ο σκοπός του ταξιδιού τους. Βεβαίως οι πέντε ώρες δεν είναι καλό από αυτήν την άποψη στα τεχνικά θέματα ε, να, βεβαίως, ε, λέμε ως πρόφαση ότι έχουμε τεχνικό πρόβλημα, υπεράριθμες κρατήσεις, αν έχετε μια οικογενική κατάσταση, άμα έρχεται από, ε, από, διά, από διάφορα αεροδρόμια και αν ένα άτομο δεν μπει στο αεροπλάνο, νομίζω ότι επηρεάζεται όλη η ομάδα, όλη η οικογένεια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα αυτό για τις υπεράριθμες κρατήσεις. Η κυρία Σανάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Αυτή, κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας μάθαμε πολλά. Ήθελα όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις έκτακτες περιστάσεις. Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το θέμα, καθώς και το θέμα της μίας μόνο χειραποσκευής. Ως προς τις ανταποκρίσεις και την πληροφόρηση που δίδεται στους επιβάτες, πράγματι πρέπει η πληροφόρηση αυτή να δίδεται πριν φτάσει ο επιβάτης στο αεροδρόμιο. Ε, πολλοί επιβάτες έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση όταν ενημερώνονται μόνο όταν και αν φτάσουν στο αεροδρόμιο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά. Θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια μου διότι δεν σημειώσαμε καθόλου προόδο στο θέμα της αφαιρεγγιότητας των αερομεταφορέων με το σύστημα του, του Collective Redress. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη ε, καταφέρει ε, να ολοκληρώσουμε αυτό το στάδιο της κατάρτισης των δικαιωμάτων των επιβατών και τώρα είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Η πρόταση αυτή έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Η κρίση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη για να ε, οπισθοχωρήσουμε. Αντιθέτως, θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε όλους τους κλάδους και αυτόν τον κλάδο το συγκεκριμένο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τα δικαιώματα των επιβατών και λαμβάνοντας υπόψη όλες μας τις ε, ε, δυνατότητες. Όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε δεν θα πρέπει να ε, πάμε προς τα πίσω, αντιθέτως, να πάμε προς τα μπροστά. Όλοι ταξιδεύουμε, οι περισσότεροι από εμά ε, ταξιδεύουμε, είμαστε επιβάτες ε, των αεροπλάνων, παίρνουμε πολύ συχνά αεροπλάνο για να έρθουμε στις Βρυξέλλες ή για να πάμε στο Στρασβούργο και έχουμε προσωπική εμπειρία και καλή και κακή ε, για το τι συμβαίνει στις διάφορες περιστάσεις και καταστάσεις τις οποίες δεν θα χαρακτήριζα καθόλου έκτακτες, μάλιστα αρκετά συνηθισμένες ενδεχομένως πολλές φορές είναι πράγματα που γίνονται. Πολλές φορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έκτακτα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αερομεταφορείς, ορισμένοι αερομεταφορείς τουλάχιστον, ε, καταχρώνται αυτή τη δυνατότητα που έχουν να μην φέρονται σωστά στους ε, επιβάτες. Υπό αυτή την έννοια η πρόταση της Κομισιόν προσπαθεί να δώσει λύσεις. Ε, Υπάρχει κρίση, ταλανίζονται οι εταιρείε, δεν είμαστε τρελοί εδώ στο Κοινοβούλιο, το γνωρίζουμε αυτό. Ε, όμως ένα χρόνο πριν από τις εκλογές δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και να αμελήσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Και οι ίδιε οι εταιρείε έχουν υποφεληθεί από ε, την ευρεία ε, χρήση των πτήσεων. Οι Ευρωπαίοι πολίτε όλο και περισσότερο ταξιδεύουν με αεροπλάνο για λόγου επαγγελματικού, για λόγου ψυχαγωγίας, για διακοπέ. Καλό είναι λοιπόν στην παρούσα κρίση να ε, κάνουμε βήματα προς τα μπροστά και να βελτιώσουμε την ποιότητα. Είναι αναγκαίο να τεθεί και το θέμα της κατάρτισης του προσωπικού για να μην έχουμε άσχημη συμπεριφορά και άσχημη αντιμετώπιση από πλευράς προσωπικού, κυρίως όσον αφορά στις εταιρείε χαμηλού κόστους και θα πρέπει να καθοριστούν ξεκάθαρα οι ευθύνες αερολιμένων και αερομεταφορέων, αλλά και επιβατών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά θέματα έχουν θυγεί. Το θέμα των υπεράριθμων πτήσεων όμως με απασχολεί ιδιαιτέρως. Αγοράζει κανείς έναν άβλο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρεί και να εφαρμόζει τις ρήτρες της σύμβασης. Διευκρινίζονται δηλαδή οι δυνατότητες ακύρωσης του εισιτηρίου από πλευράς επιβάτη. Δεν υπάρχει ρήτρα που να, να δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να ξαναπαίρνει ένα εισιτήριο που έχει ήδη ε, πωλήσει. Εγώ νομίζω ότι αυτό δίνει λαβή για ποινική ευθύνη δεν θα πρέπει μόνο να απαγορεύεται, αλλά να υπάρχουν κυρώσεις γι' αυτό, θα πρέπει να ποινικοποιείται. Είναι πραγματικό το ζήτημα, είναι αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, το γεγον... κανείς έμπορος δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν έχει πουλήσει ένα εισιτήριο να το ξαναπουλάει και σε άλλον ουσιαστικά. Δεν είναι ρήτρα τα να είναι γεμάτες, γεμάτα τα καθίσματα ή το θέμα της χρήσης των ΣΛΑΟΤΟ, όλα αυτά μπορούν να δώσουν λαβή για λύση της σύμβασης μεταξύ εταιρεία και επιβάτη. Θέλω να είναι εξαιρετικά δεσμευτική η διατύπωσή μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και εγώ, από τη δική μου πλευρά, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Αυτό το οποίο είναι σαφές σήμερα είναι το εξής. Ο... κανονισμό αυτό τον ε, ερμηνεύουν διαφορετικά οι διάφοροι αερομεταφορείς και έτσι είναι σαφής η ανάγκη αναθεώρησης και μεταρρύθμισης. Άλλες εταιρείε ε, συμμορφούνται με τους κανόνες, άλλες ε, λειτουργούν διαφορετικά. Αυτό είναι ε, που κυρίως ενοχλεί τα μέλη. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε. Και υπάρχει και το θέμα της που έθεσε η κυρία Γιάλα Σέντερ, η πλήρης άγνοια που επικρατεί ε, στα αεροδρόμια, όχι μόνο ε, από πλευράς προσωπικού αεροπορικών εταιριών, αλλά και από πλευράς προσωπικού ε, υπηρεσιών εδάφους, handling κτλ. Για το τι είναι αυτός ο κανονισμός και τι προβλέπει. θα ξέρετε αυτή την ιστορία που ε, με έστειλαν στο κέντρο ε, αστυνομικό ε, του Μάντσεστερ πολύ απλά γιατί έθεσα μια ερώτηση για το ποια είναι τα δικαιώματά μου ως επιβάτης. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, τέτοιου είδους περιστατικά ε, μας δημιουργούν ε, συναισθήματα πολύ αρνητικά, όχι μόνο σε μένα αλλά και στα υπόλοιπα μέλη. Εγώ λαμβάνω και πάρα πολλές καταγγελίες και παράπονα από την εκλογική μου περιφέρεια. Και εκεί δεν έχουμε διετερικές συνεργασίες και συμφωνίες. Έχουμε ταξίδι από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Πτήσεις, τσάρτερ σε μεγάλο βαθμό, ναυλωμένες, αλλά εν πάση πτώση έτσι έχει το πράγμα. Συμφωνώ με την κυρία Φώστερ. Εάν εντάσσονται αυτά στο, στην οδηγία για τα τουριστικά πακέτα, τότε δεν θα πρέπει να παίρνει κανείς διπλή αποζημίωση και για το τουριστικό πακέτο αλλά και για πτήση. Το, δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Αυτό Τόσο τομέα τομέας είναι που πλήττεται περισσότερο. Εκεί πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό. Καταλαβαίνω ε, το θέμα της ανωτέρας βίας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θεωρείτε ότι η Κομισιόν έχει σημειώσει πρόοδο, ωστόσο σε άλλα ζητήματα η Κομισιόν δεν έχει, καθόλου, ε, δεν έχει σημειώσει καθόλου πρόοδο. Περιμένουμε λοιπόν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη συζήτηση που ε, θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Να δώσω στην Κομισιόν το λόγο για τις καταληκτικές της παρατηρήσεις και μετά να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Κόλσον, έχετε κάτι να πείτε. Όχι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ωραία, πολύ σόφρον αν με επιτρέπετε. Ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον απόγευμα με την συμβολή όλων και νομίζω ότι ήδη εξαγάγατε τα σωστά συμπεράσματα. Εγώ στην εισαγωγή μου ανέφερα ορισμένα θέματα Δεν ξέρω βέβαια τώρα σε ποια σημεία πρέπει κυρίως να επικεντρωθούμε, αλλά νομίζω ότι έθιξα όσα ήθελα στην εισαγωγή και για μένα δεν πάει αρκετά μακριά σε ορισμένα ζητήματα. Υποστηρίζω αυτά που είπε η συνάδελφος Ζαλανόβα για την πτώχευση, πρέπει να υπάρξουν ε, πιο δεσμευτικές ε, ρυθμίσεις και για τους ορισμούς, τους ορισμούς, της ε, αρμοδιότητες, εδώ υπάρχουν πολλά που πρέπει να λύσουμε μεταξύ αεροδρομίων, εταιριών και ποιος είναι υπεύθυνο για ποια πληροφόρηση. Και ο ορισμός των ατόμων με ειδικέ ανάγκες ή με περιορισμένη κινητικότητα και εδώ χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Ορισμένα σημεία τα καλωσορίσαμε και εγώ το κάνω ε, σχέδια για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ε, πολύ βασικό. Τώρα πώς ακριβώς ε, λεπτομερώς θα εκπονηθούν, πρέπει ακόμη να καταρτιστεί. Συμφωνώ με διάφορους ομιλητές ότι αυτό το όριο πέντε ωρών σε πολλές περιπτώσεις είναι επιδίνωση. Χειρότερο από ό,τι προηγουμένως. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νομολογία η Κομισιόν δεν την αγνοεί βεβαίω, αλλά επεχείρησε να δει μόνο νομικά, να ερμηνεύσει μόνο νομικά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει όμως να ληφθούν αυτές οι, αποστάσεις, οι αποφάσεις πιο συγκεκριμένα υπόψη και για τις ε, χειραποσκευές πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Γενικά Είμαι ευχαριστημένος και από τη συνεργασία με τους ηγητές άκουσα πολύ ενδιαφέροντα ε, θέματα. Ευχαριστώ και την ΙΜΚΟ, ευχαριστώ για την διοργάνωση και την ε, ε, διεύθυνση της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ζόρζ λέει ο Πρόεδρος. ένα λεπτό παρακαλώ οι εκπρόσωποι που είχαν πάρει το λόγο. Ένα λεπτό καθένας. Είναι το δικαίωμα απάντησης. Είμαι δημοκράτης έτσι δεν είναι. Φόξ για τα αεροδρόμια ένα λεπτό. Αυτό που είπε η κυρία Βερνιό θέλω να αναφέρω, η ανάγκη να υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης ότι είναι θετικό και να καθορίσουμε τους κανόνες και τις ευθύνες εντός των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για να μην υπάρχει σύγχυση για τους επιβάτες ποιος είναι υπεύθυνο για ποιο δικαίωμά τους και να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε έχουν έναν ε, εκπρόσωπο επιτόπου για να ασχοληθεί με τους επιβάτες σε περιπτώσεις προβλημάτων και ευχαριστώ. Κυρία Ντεσμέτ. Ένα μόνο. Πολλές ανησυχίες άκουσα για τις πέντε ώρες ε, ως πρώτο κατόφλι ενεργοποίησης. Τα κατόφλια είναι αναγκαία για τις εταιρείες για να αντιμετωπίσουν την καθυστέρηση και για να προσπαθήσουν να διεξαχθεί όντως η πτήση. Πέντε ώρες. Στον κανονισμό αυτό θεωρείται το κατόφλι για την μακροχρόνια καθυστέρηση από το οποίο και μετά έχει δικαίωμα αποζημίωση ο επιβάτης. Είναι λογικό λοιπόν. Επιμένω ότι είναι προς το συμφέρον των επιβατών οι εταιρείε να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το αίτιο του προβλήματος και να μην ακυρώνουν τις πτήσεις. Δεν σημαίνει πως δεν θα φροντίσουμε για τους επιβάτες μας, δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε να πληρώσουμε αποζημίωση. Επιπλέον από την καθυστερημένη πτήση. Ευχαριστώ. Μαγναμάρα, ένα λεπτό. Όχι, ευχαριστώ. Χάνλον. Λίγα παραπάνω για αυτά που, είπαμε, που είπε και η Άτα. Είμαστε υπέρ της εξήγησης, αλλά έκανε ερώτηση η κυρία Πάκε από την εταιρεία καταναλωτών γιατί υπάρχει αυτή η επιδίνωση σε σχέση με τις συνθήκες αποζημίωσης για τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Μα νομίζω ότι είναι αυτονόητη απάντηση. Η εταιρεία, εάν πρόκειται να δώσει αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις και δεν προλαβαίνει να βρει εναλλακτική λύση, έχει κάθε συμφέρον να ακυρώσει την πτήση, ούτως ώστε να περιορίσει το κόστος. από τι απαιτήσει αποζημίωση από όλου του άλλου. Αυτό όμω δεν είναι προ το συμφέρον των καταναλωτών που θέλουν να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Άρα το χειρότερο για αυτού είναι να ακούσουν ότι ακυρώθηκε όχι απλώ καθυστέρησε η πτήση του. Δύο θέματα. Ο πελάτη είναι στην καρδιά τη επιχείρησή μα. Αν δεν του αντιμετωπίζουμε σωστά δεν θα έχουμε επιβάτε. Προσπαθούμε λοιπόν πάντα να σεβαστούμε του πελάτε και τα δικαιώματά του. Θα ήταν κρίμα αυτή η συζήτηση για να γίνει τελικά συζήτηση αντιπαράθεσης μεταξύ του κλάδου και των επιβατών. Όχι. Όσοι επιβάτες έχουν πρόβλημα, βεβαίως ε, πρέπει να τύχουν σωστής αντιμετώπισης, αλλά για όλους τους επιβάτες θα μειωθούν τα δικαιώματα εάν το καθεστώς που επιβληθεί είναι ιδιαίτερα ε, βαρύ. Επίσης, Υπάρχει κάποια παρανόηση. Δικαίωμα αποζημιώση. Μπορεί να θεωρείται από ορισμένου ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Όχι. Είναι το κατώτατο όριο στο οποίο έχει δικαίωμα ένας επιβάτης. Εάν ο επιβάτης έχει επιπλέον βλάβη υποστή λόγω τη καθυστέρηση, έχει και συμπληρωματικά δικαιώματα για να ζητήσει περαιτέρω αποζημίωση είτε μέσω της Σύμβασης Μοντρεάλ είτε μέσω της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια. Ναι, ήθελα απλώς να αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα της αφαιρεγγιότητας ε, επιβολής ε, των νόμων και τήρησης των αποφάσεων του δικαστηρίου. Να υπάρχει με ίσους όρους ανταγωνισμό και θα πρέπει όλοι να παίζουν το παιχνίδι με τους ίδιους κανόνες. Και ε, κυρία Πάχλ, τελευταία, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω σύντομα σε ένα σημείο που ε, αναφέρθηκε, η κυρία Φώστερ που ασχολείται με την καρδιά του θέματος, διότι είπε ότι οι υποχρεώσεις είναι και ε, στις δύο μεριές των συμβαλωμένων. Έχουν υποχρεώσει και οι αερομεταφορείς και οι επιβάτες, διότι πολύ συχνά οι αερομεταφορείς δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και νομίζω ότι μας εκπλήσει ότι είναι ένας τομέας που δεν ακολουθεί τα ίδια πρότυπα ε, δικαιοσύνης όπως άλλοι οικονομικοί τομείς. Και όπως εξήγησα προηγουμένως υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει νομολογία, πολλές αποφάσεις δικαστηρίων και πάρα πολλοί όροι συμβατικοί είναι άδικοι και χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς και συνιστώνται από την ΙΑΤΑ και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είχε, έχει πει σχετικά με τη ρήτρα της μη εμφάνισης. Βεβαίως η εφαρμογή είναι σημαντική αλλά τώρα είναι ευκαιρία ε, οι ουσιαστικοί κανόνες να γίνουν σωστοί και δίκαιοι και να βλέπουμε πώς μπορούν να επιβληθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξοδέψαμε πολύ ε, χρόνο για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα, αλλά βεβαίως πρέπει να ασχοληθούμε με την επιβολή ε, των κανόνων, την εφαρμογή από τους ε, τομείς που πρέπει ε, να εξεταστούν, να εξεταστεί ο ρόλος των εθνικών οργάνων επιβολής των νόμων. Σας ευχαριστώ όλους που εκθέσατε τις απόψεις εδώ στην Επιτροπή. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, προθεσμία για τροπολογίες στην εισήγηση αυτή 3 ε, Οκτωβρίου με εξέταση των τροπολογιών στην συνάντηση της 5ης Νοεμβρίου και ψηφοφορία στις 14 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Ολομέλεια, δεν ξέρουμε πότε. Ελπίζουμε να φτάσουμε στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο με την εισήγηση αυτή του 2014. Για τα μέλη, η εξέταση του σχεδίου εισήγησης ε, θα είναι στις 16-17 Σεπτεμβρίου στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον εισηγητή, τους Όδης εισηγητές για την εργασία τους και τώρα ε, και κλεισμένων των ε, θυρών θα ασχοληθούμε με την, τους τριμερείς διαλόγους.